αφορά τι τρίτε χώρε, αναπτυσσόμενε χώρε και πρέπει να τι βοηθήσουμε. Είναι σωστό. Thank you. Σας ευχαριστώ και θα ήθελα να επεκτείνω τις ευχαριστίες μου και σε όλους τους άλλους που συνεργάστηκαν έτσι ώστε να καταρτήσουμε αυτό το κείμενο. Συμφωνώ, το κείμενο που έχουμε μπροστά μας αποτελεί μια καλή βάση για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε. Ταυτόχρονα πιστεύω θα ήταν χρήσιμο να επιστήσουμε την ιδιαίτερη προσοχή όλων στο πώς μπορούμε να κάνουμε πιο ξεκάθαρο και σαφές το κείμενο. Για να μην δώσουμε την εντύπωση ότι επειδή μιλάμε για τις δικές μας ευθύνες και για τη μείωση, δεν καταλαβαίνουμε το ότι είναι εξίσου σημαντικό να υπάρξει ισχυρή πολιτική και φιλόδοξη συμφωνία όσον αφορά την προσαρμογή. Όσον αφορά το επίπεδο φιλοδοξία, συμφωνώ με του συναδέλφου που πήραν το λόγο προηγουμένω. Πραγματικά πρέπει να μιλήσουμε για 40% και όχι να παραπέμπουμε σε ένα ανώτατο όριο 25%. Ε, όσον αφορά τη μείωση. Ταυτόχρονα πιστεύω ότι το ποσό της χρηματοδότησης, ιδιαίτερα όταν αναφέρουμε στην παράγραφο 8 ένα συγκεκριμένο αριθμό, αυτό το ποσό είναι πολύ χαμηλό. Αν θέλουμε να αναφέρουμε συγκεκριμένα ποσά, πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι όσον αφορά ε, τα χρήματα τα οποία θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε. Και για τη χρηματοδότηση. Δεν θα πρέπει να μιλάμε μόνο Ε, για τα χρήματα, αλλά και για το μηχανισμό. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ε, ιδιαίτερα αν συμπεριλάβουμε και ορισμένε ιδέε από την Επιτροπή Ανάπτυξη. Να κάνουμε λοιπόν, ε, να, να αναλάβουμε συγκεκριμένη δέσμευση και από τη δική μα σκοπιά, για να δούμε γιατί ακριβώ μιλάμε και τι πρέπει να πούμε στο Συμβούλιο. Πιστεύουμε ότι οι αναπτυσσόμενε χώρε θα πρέπει να πούν πολύ περισσότερα και όσον αφορά το μηχανισμό διανομή και κατανομή των χρημάτων. Ταυτόχρονα πιστεύω ότι πρέπει να ενισχύσουμε αυτά τα οποία αναφέρουμε για την προσέγγιση μα προ την τεχνολογική συνεργασία, μεταφορά τεχνολογία και όσον αφορά την αποψήλωση των δασών, ίσω θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για μηδενική ε, αποψήλωση, ακριβώς για να ενισχύσουμε τις δικές μας απόψεις και να πούμε τι ακριβώς θέλουμε. Συμφωνώ επίσης ότι στο κείμενο θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε σαφώς ότι από τη μια μεριά τονίζουμε ότι μείωση των εκπομπών πρέπει να γίνει στις εκβιομηχανοποιημένες χώρες και να μην ε, γίνεται κάπου αλλού, αλλά ταυτόχρονα όμως πρέπει να βοηθήσουμε και τις αναπτυσσόμενες χώρες. Ε, αν θέλουμε και οι χώρες αυτές να συμβάλλουν προς την κατεύθυνση που ελπίζουμε και εμείς να συμβάλλουν με τις δικές τους δεσμεύσεις, έτσι ώστε να υπάρξει μια διεθνή συμφωνία. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω και εγώ όλους τους συμμετέχοντες για την ποιότητα του ψηφίσματος. Και να πω εδώ ότι εμείς ως ευρωβουλευτές εκπροσωπούμε τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο σε 50 χώρες του κόσμου και στην Ευρωπαϊκή Ένωση έγινε μια διάσκεψη συνεννητική όπου Σύνεδροι από διάφορες χώρες ε, συζήτησαν για την κλιματική αλλαγή και για τις ε, απαιτήσει που υπάρχουν. Είχαμε εκπροσώπους ε, από χώρες BRIC, από χώρες αναπτυγμένες και από όλες τις υπόλοιπες χώρες. Τα αποτελέσματα μπορείτε να τα βρείτε στο διαδίκτυο, θα σας δώσω τους σχετικούς συνδέσμους. Και αυτό που βλέπουμε είναι ότι πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα φιλόδοξοι είναι προφανές ότι το θέμα είναι επίγον για 80% των κατοίκων των νότιων χωρών και 45% μόνο των χωρών του Βορρά. Δηλαδή στις πλούσιες χώρες έχουμε πολύ λανθασμένη εντύπωση. Επίσης, περίπου 60% των ε, συμμετεχόντων θεωρούσαν ότι θα πρέπει η προσπάθειά μας να είναι 25-40% και παραπάνω. Άρα το 25% είναι πολύ χαμηλό σε σχέση με αυτό που αναμένει ο πληθυσμός από εμάς. Και ένα τρίτο θέμα, οι χώρες του Νότου ακόμη και οι λιγότερο προηγμένες είναι διατεθειμένες να προσπαθήσουν να συνεισφέρουν στον αγώνα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Μόνο 16% διαφωνούσε με αυτή την προσέγγιση. Και επίσης να πω ότι οι χώρες BRIC και οι χώρες του Νότου γενικά ήταν πολύ πιο θετικές από τους συμμετέχοντες από χώρες του Βορρά και να πω ότι σε αυτή τη διάσκεψη συμμετείχαν ε, άτομα από διάφορους επαγγελματικούς τομείς, οργανώθηκε από δανούς. Είχαμε λοιπόν ένα καλό δείγμα που μας έδειξε ποιες είναι οι προσδοκίες του παγκόσμιου πληθυσμού και του ευρωπαϊκού πληθυσμού. Οπότε εμείς που εκπροσωπούμε τον ευρωπαϊκό πληθυσμό πρέπει να τους ακούσουμε αυτούς. Ένα εμείς και δύο οι Αμερικανοί. Και πρέπει οπωσδήποτε να προσπαθήσουμε να δεσμευτούν και οι Αμερικανοί. Είπατε κύριε Πρόεδρε ότι τέλειο Οκτωβρίου θα πάει μία αντιπροσωπεία στις Ηνωμένε Πολιτείε. Θα ήταν σημαντικό να υπάρξει μία συνάντηση με κοινοβουλευτικούς στην Αμερική. Και επίσης θα έπρεπε να δημιουργηθούν έστω και μέσω διαδικτύου σύνδεσμοι επικοινωνίας μεταξύ Αμερικανών και Ευρωπαίων πολιτών. Αυτό που είδαμε ήταν ότι οι Αμερικανοί που συμμετείχαν στην εκδήλωση στην οποία ανέφερα ήταν ιδιαίτερα θετικοί, πιο θετικοί και από την κυβέρνηση Ομπάμα όσον αφορά τη λήψη μέτρων και μάλιστα λήψη δεσμευτικών και επεληθεύσιμων μέτρων. Άρα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να απευθυνθούμε απευθείας στον αμερικανικό πληθυσμό και με αυτό που θα πρέπει να ασχοληθούμε στο μέλλον. Και τέλος, όσον αφορά τη χρηματοδότηση, το ανέφεραν και οι συνάδελφοι. Πρέπει να υπάρξει δημόσιος και διεθνής, ε, δημόσια και διεθνής χρηματοδότηση. Δεν ξέρω τι θα βρούμε, φόρος για τις μεταφορές, φόρος Τόμπιν, φόρος ε, που θα προκύπτει από την εμπορία των εκπομπών. Πάντως κάτι πρέπει να βρεθεί για τη χρηματοδότηση της αντιμετώπισης της αλλαγής στις χώρες του Νότου. Και πρέπει να υπάρξει και προσαρμογή. Τι εννοώ προσαρμογή. Προσαρμογή της συμπεριφοράς μας προκειμένου να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή. Παράλληλα όμως προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Και όσο πιο γρήγορα κινητοποιήσουμε τους συμπολίτες μας με κατάλληλα μέτρα προκειμένου να μάθουν ποιε θα είναι οι συνέπειες για τη ζωή τους από τις ήδη υπάρχουσες κλιματικές αλλαγές, τόσο πιο γρήγορα θα μπορέσουμε να έχουμε αυτά αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Μία εκστατεία από το ίντερνετ των Ευρωπαίων προς την κατεύθυνση των Αμερικανών γερουσιαστών Ξέρω ότι οι Αμερικανοί έχουν εστιάσει την προσοχή τους περισσότερο στην Κίνα και όχι στην Ευρώπη. Δεν τους νοιάζει τόσο η Ευρώπη, αλλά περισσότερο τι κάνει η Κίνα ή τι δεν κάνει η Κίνα. Αυτό είναι ένα πρόσθετο πρόβλημα ότι κοιτάνε αλλού οι Αμερικανοί από εκεί που εμείς θέλουμε να τους στρέψουμε την προσοχή. Δεν είμαστε τόσο ορατοί και τόσο σημαντικοί για τους Αμερικανούς όπως οι Κινέζοι. <clears throat> και αυτό είναι ένα πρόσθετο πρόβλημα. Ε, Σλούτερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ την ε, προηγούμενη Δευτέρα εκπροσωπούσα την Επιτροπή μας στη Στοκχόλμη μέσα στην ε, ε <coughs> διάσκεψη αυτή που αφορούσε την ανάπτυξη και τα προβλήματα της ε, προστασίας του περιβάλλοντος. Θυμίζω το ψήφισμα του Απρίλιου, στο οποίο είχαμε πολύ καλές διατυπώσεις για το ζήτημα αυτό της ε, εξασφάλισης των δικαιωμάτων των λαών του τρίτου κόσμου, ότι εμείς ως εκπρόσωποι του πρώτου κόσμου δεν πρέπει να ασχολούμεθα μονάχα με τα δικά μα ευρωπαϊκά δάση. Και επομένως, εάν θέλουμε πραγματικά να είμαστε ε, αξιόπιστοι σε σχέση με το στόχο αυτό της μη αύξησης πάνω από το 2%, δύο βαθμούς μάλλον και θέλουμε να έχουμε μια πιθανότητα τουλάχιστον 50% να επιτύχουμε το στόχο αυτό, είναι απαραίτητο να τονίσουμε τη σημασία αυτού του στόχου και να έχουμε τα 300 δισεκατομμύρια ως το ποσό το οποίο πρέπει να είναι χρηματοδότηση της ε, προστασίας του κλίματος. Αυτό όμως θα πρέπει να το θέσουμε σε ένα πλαίσιο σύγκρισης με άλλες χρηματοδοτήσεις. Και επίσης θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι μειώσεις των εκπομπών αερίων του, θερμο, του θερμοκηπίου που μπορούμε να επιτύχουμε και σε άλλες χώρες. Εμείς λέμε είμαστε έτοιμοι να φτάσουμε στο 40% αλλά θα είναι χρήσιμο να πούμε ότι είμαστε και έτοιμοι να χρηματοδοτήσουμε άλλες χώρες για να φτάσουν και αυτές σε αντίστοιχες μειώσεις των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στην πολιτική μα. Είναι γεγονό ότι η Κίνα είναι σημαντική. Είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να φέρουμε την Κίνα στο δικό μα στρατόπεδο. Και είναι απαραίτητο να τονίσουμε την αξία των προϊόντων τα οποία έχουν μεγαλύτερη ενεργητική αποδοτικότητα και τη μεγαλύτερη χρήση της, ε, ε, των εναλλακτικών ενεργειών, όπως παραγματικά η δημιουργία εγκαταστάσεων φωτο, ε, φωτοβολταϊκής ενέργειας. Υπάρχουν όμως πολλές ακόμα πολλά εμπόδια για να μπορέσουμε εμείς να πουλήσουμε τα προϊόντα μας στις χώρες του τρίτου κόσμου και ιδίως στην Κίνα. Είναι απαραίτητο λοιπόν να αναπτύξουμε μια αγορά παγκόσμια για τα προϊόντα ανανεώσιμης ενέργειας. Επομένως αυτό θα ήταν χρήσιμο να μπορέσει να μας οδηγήσει σε μια σημαντική μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρωπο. Νομίζω ότι εμεί θα πρέπει να τονίσουμε το στόχο του 30% γιατί είναι θετικό και για το περιβάλλον και για την ευρωπαϊκή βιομηχανία προϊόντων ανανεώσιμη ενέργεια. Και στη συνέχεια έχουμε τις ε, συμφωνίες που έχουμε ήδη συνάψει. Η Ισπανία ήδη εκπέμπει 35% περισσότερες, περισσότερα αέρια θερμοκηπίας από ό,τι προβλέπεται στο Κιώτο, στον πρωτόκολλο του Κιώτο. Θεωρείτε όμως ότι μπορέσει η Ισπανία να πετύχει το στόχο που έχουμε θέσει μέχρι το 2020. Μάλλον όχι. Επομένως θα πρέπει να αναλάβουμε την ευθύνη του να πράξουμε κάτι μέσα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλιώς δεν θα μπορέσει να επιτευχθεί ποτέ αυτός ο στόχος σε ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και υπάρχουν άλλες χώρες οι οποίες απέχουν 10% από τους στόχους του Κιώτο. Επομένως, ενώπιον τη Κοπεχάγη, εμεί θα πρέπει να αναλάβουμε και περαιτέρω δεσμεύσει για να μπορέσουμε να πείσουμε και χώρε όπως η Ιαπωνία και η Κίνα. Είναι απαραίτητο να εξασφαλίσουμε τη δική μας αξιοπιστία. Και αν αυτό απαιτεί και αλλαγέ του τρόπου ζωής. Ναι, υπάρχουν ενδιαφέρουσες προτάσεις, Παραδείγματο χάρη μια μείωση του χρόνου εργασία. Αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει την ε, επίτευξη των στόχων του, της κλιματικής αλλαγής. Μια μείωση λοιπόν του χρόνου εργασίας, ιδίως αν αυτό θα ανακουφίσει και πάρα πολλά άτομα τα οποία αυτή τη στιγμή είναι άνεργα, αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ τα πράγματα. Ίσως λοιπόν θα πρέπει να εξετάσουμε και πάλι αυτές τις δυνατότητες και να λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι πάρα πολλοί εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν μια τεράστια κόπωση, ένα burnout μετά από πολλά χρόνια εργασίας. Λοιπόν, μια αλλαγή του χρόνου εργασία, το να δώσουμε στου εργαζόμενου περισσότερο χρόνο για τι οικογένειε και τα παιδιά του, αυτό θα είναι θετικό και για το κλίμα. Κυρία Γκροστέτ, έχετε το λόγο. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα να πω συναδέλφου μα που ήρθαν τώρα στο Κοινοβούλιο ότι αυτή τη στιγμή δεν ε, Πρωτό τα ζητήματα αυτά. Εδώ και πολλά χρόνια εργαστήκαμε, και το ξέρουν οι παλιοί συνάδελφοι, εργαστήκαμε σε αυτό το θέμα και την αντιμετώπιση του προβλήματο τη κλιματική αλλαγή. Σα υπενθυμίζω την προσωρινή Επιτροπή για το Κλίμα με ευθύνη του συναδέλφου μα, του κυρίου Φλόρεντ. Όταν βλέπω σήμερα, ή μάλλον ακούω σήμερα όλα αυτά μου δημιουργείται η εντύπωση ότι εδώ υπερθεματίζουμε όλοι. Ποιος θα πει περισσότερα, 30, 40, 100, 50%. Λέει κάποιο. Πού είναι η αξιοπιστία σε όλα αυτά, Πού βρίσκεται ο ρεαλισμός. Πραγματικά έχω την εντύπωση ότι ονειρεύομαι. Ε, είναι φοβερά όλα αυτά. Είμαστε ε, μέλη του Κοινοβουλίου, πρέπει να είμαστε σοβαροί σε αυτά τα οποία προτείνουμε και να λάβουμε υπόψη όλα τα ε, δεδομένα που έχουν βεβαίω να κάνουν με την κλιματική αλλαγή, αλλά και τα οικονομικά δεδομένα και τους εταίρους μας. Ε, ε, γιατί ξέρουμε εκτό τη Κοπεχάγη ότι θα είναι δύσκολα. Η τελευταία συνεδρίαση στη ΣΥΠΑ έδειξε ότι δεν πρέπει να θεωρούμε καθόλου κεκτημένο αυτό το θέμα. Και μάλιστα εγώ αισθάνομαι μάλλον απεσιοδοξία. Η Ευρώπη θέλει να είναι υποδειγματική. Βεβαίω, έχουμε κάθε δίκιο. Αλλά ε, αυτό δεν σημαίνει ότι ε, εμείς ε, θα προσπαθούμε διαρκώς να είμαστε μπροστά από τους άλλους, χάνοντας όμως την αξιοπιστία μας γιατί διαφορετικά δεν θα πείσουμε κανέναν. Ακούω τον πρόεδρο και έχει δίκιο που το λέει και το υπεθυμίζει. ότι οι έχουν το βλέμμα του στραμμένο στην Κίνα και μάλλον μηδίαμα τους προκαλεί η Ευρώπη. Άρα πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα. Έχουμε να λάβει συγκεκριμένε δεσμεύσει για τη Κοπεχάγη. Πρέπει να εμείνουμε σε αυτέ τι δεσμεύσει και να μην ξεπεράσουμε. Να μην ξεπεράσουμε. Εάν τηρήσουμε τις υποσχέσεις μας, τότε πραγματικά θα έχουμε σημειώσει πρόοδο. Και τότε έχουμε το καθήκον ε, να προχωρήσουμε περισσότερο. Γιατί εγώ είμαι πεπισμένη ότι πρέπει να προχωρήσουμε με στάδια. Να θέλουμε από την αρχή ε, να πάμε πολύ μακριά. 15 χρόνια μέσα σε αυτό το κοινοβούλιο. Το ξέρω από την πείρα μου. Αν ε, βάζουμε τον πύχη πολύ ψηλά, έτσι κι αλλιώ δεν πρόκειται να φτάσουμε πουθενά. Και θα αποτύχουμε. Δεν είμαι σίγουρη λοιπόν ότι αυτό είναι το καλό μέσον γιατί πρέπει να πείσουμε τους εταίρους μας για να καταβάλουμε όλη κάθε προσπάθεια έτσι ώστε να περιορίσουμε την αύξηση σε αυτούς τους δύο βαθμούς. Να είμαστε με στο στόχο του 2%. Συμφωνούμε. Αλλά εγώ θα ήθελα να σας πω το εξής. Όταν μιλάμε για μεταφορά τεχνολογίας από τις βιομηχανημένες χώρες, βεβαίως πρέπει να, ε, να δώσουμε το καλό παράδειγμα. Πρέπει να συμμετάσχουμε σε αυτή την προσπάθεια και να μεταφέρουμε την τεχνολογική μας ε, πρόοδο και στις υπόλοιπε χώρε. Αλλά πρέπει οπωσδήποτε να σεβαστούμε και το θέμα, τα θέματα, για παράδειγμα, προστασία πνευματική ιδιοκτησία. Είναι θεμελιώδε αυτό το σημείο. Και κάτι άλλο. Να μην ε, ε, να καταλάβουμε ότι αν τελικά δεν καταφέρουμε να πείσουμε τους Αμερικανούς, γιατί υπάρχουν ανησυχίες, τότε θα πούμε ότι δεν έχουμε συμφωνία ή ότι η συμφωνία δεν είναι ικανοποιητική. Μα κοιτάξτε, τότε πρέπει να, υπάρξει, να προτείνει η Επιτροπή Μηχανισμό Προσαρμογή στα Σύνορα, ε, που ε, να λαμβάνει υπόψη τι ποσοστώσει εκπομπών αερίου θερμοκηπίου ε, από το 2013 μέχρι το 2020. Έτσι ώστε, πώ να το πω, να υπάρξει μια κάποια εναρμόνιση των όρων του ανταγωνισμού με τι αναπτυγμένε χώρε που δεν θα έχουν τηρήσει τη δέσμευσή τους ε, για μείωση όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εφιστώ την προσοχή όλων. Προσοχή. Ο στόχος είναι κοινό. Όλοι θέλουμε να κάνουμε κάθε προσπάθεια για να καταπολεμήσουμε την αλλαγή του κλίματος. Σας παρακαλώ όμως. Ας επιδείξουμε ρεαλισμό, ας προχωρήσουμε με ε, στάδια. Βεβαίως να ασκήσουμε πίεση στους ε, Αμερικανούς και σε όλους τους εταίρους έτσι ώστε να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους. Αλλά προτείνοντας μείον 40%, μείον 50% πιστεύετε ότι θα πετύχουμε το στόχο μας, αντίθετα χάνουμε αξιοπιστία. Αυτά ήθελα να πω. Νομίζω ότι πραγματικά πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι μέχρι την Κοπεχάγη πρέπει να πείσουμε τους Αμερικανούς εταίρους μας αλλά ε, κυρίως αυτό που θέλω να πω είναι να μην βάζουμε εμπόδια στη δική μας την πορεία. Ευχαριστούμε η κυρία Ντάγμαντ ε, Ροτμπέρεντ για θέμα τάξη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Είναι πράγματι ένα θέμα διαδικαστικό Θέλω να υπενθυμίσω λοιπόν τη σωστή διαδικασία. Έχουμε να συνεδριάσουμε εδώ όλη μέρα. Ξέρουμε αυτό το χώρο, ξέρουμε την ακουστική της αίθουσα της ε, Ολομέλειας. Εγώ βγαίνω με ποροκεφάλους κάθε φορά. Ακούμε όλους τους ομιλητές με ηχό. Είμαστε υποχρεωμένοι να ακούμε μόνο από τα ακουστικά, ακόμα και για τις γλώσσε που ακούμε. Και είναι θέμα τεχνικής Ίσως θα πρέπει να εξασφαλίσουν οι τεχνικοί ότι έχουμε στον χώρο της Ολομέλειας τον την απαραίτητη ποιότητα ήχου για να μπορούμε να παρακολουθούμε τις συνεδριάσεις με έναν τρόπο ο οποίος θα είναι ικανοποιητικός. Λοιπόν, πρέπει να κάνουμε κάτι. Δεν μπορούμε να συνεχίζουμε έτσι. Είναι πάρα πολύ κουραστικό αυτό το να ακούμε κάτω από αυτές τις συνθήκες ήχου στην Ολομέλεια της ε, συνεδριάσης μας. Κυρία Πρόεδρε, τα διαβήματα αυτά έχουν γίνει ήδη στο παρελθόν χωρίς μεγάλη επιτυχία. Δεν έχει βελτιωθεί η κατάσταση της ε, ακουστικής, ούτε εσείς ούτε εμείς είμαστε τεχνικοί. Δεν μπορούμε εμείς λοιπόν να εκτιμήσουμε το, ότι, το αν επιτυχήσει ή όχι προσπάθειες των τεχνικών, μόνο αυτοί μπορούν να βελτιώσουν την άνεση με την οποία μπορούμε να παρακολουθούμε τις συζητήσεις από ηχητική πλευρά. Αυτό το οποίο θα ήθελα όμως να σας ζητήσω είναι να απομακρύνετε τα ακουστικά σας από το μικρόφωνο όταν μιλάτε για να μην υπάρχουν μικροφωνισμοί. Γιατί σίγουρα αυτοί οι μικροφωνισμοί δημιουργούν αυτή την ε, ατμόσφαιρα σύγχυσης ηχητικής η οποία είναι πράγματι ενοχλητική. Δίνω τώρα το λόγο. Δεύτερο διαδικαστικό, δεύτερη διαδικαστική παρέμβαση του κύριο Φλόρεντς. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να, να σας τονίσω ότι ίσως θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι πολλές φορές η διοίκηση του Κοινοβουλίου θεωρεί ότι εμείς είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι και αυτή η εντύπωση είναι λαθασμένη. Δεν πρέπει να υπάρχει αυτή η άποψη πιστεύω. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Αρσέντς έχει το λόγο. Thank you, Mr. President. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και εγώ συμφωνώ ότι είμαστε υπερβολικά αισιόδοξοι όσον αφορά τους στόχους μας. Δυστυχώς όμως σύντομα θα πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερα όσον αφορά τις ευθύνες του αναπτυσσόμενου κόσμου. Εμείς θα πρέπει να προσφέρουμε την χρηματοδότηση. Και αναφέρει η ανακοίνωση της Επιτροπής ότι θα πρέπει να έχουν μείωση 15 με 30% αν και αυτό δεν αναφέρεται και στο έγγραφό μας. Εν πάση περιπτώσει το έγγραφο είναι πολύ καλό και θα ήθελα να συγχαρώ όλους όσους συνεισέφεραν. Τώρα, ένα σχόλιο για αυτό που αναφέρθηκε για τη σχέση ΙΠΑ και Κίνας. Έχω ζήσει κάποιο καιρό στις Ηνωμένε Πολιτείε και θεωρώ ότι παρόλο που η κυβέρνηση της Αμερικής ασχολείται ιδιαίτερα με την Κίνα, ο πληθυσμός της Αμερικής και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις κοιτάνε κυρίως προς την Ευρώπη. Εμείς ξεκινήσαμε το διαφωτισμό στην Ευρώπη και εμείς πρέπει να είμαστε και τώρα αυτοί που θα είμαστε στην πρωτοπορία. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Ντέιβις. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Χαίρομαι που ακούω την όλη συζήτηση. Εγώ ένα πράγμα θα ήθελα να πω. Αυτό που είχαμε διαπιστώσει από τις προηγούμενες διασκέψεις ήταν μία βηματική αύξηση. Ένα-ένα βήμα κάθε χρόνο. Στην Κοπενχάγη ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να κάνουμε ένα μεγάλο βήμα προς το εμπρός και θα δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο για πιο φιλόδοξα μέτρα. Ακούσαμε από το Σουηδό Υπουργό ότι για αυτόν οι ελάχιστες προϋποθέσεις για επιτυχία στην Κοπενχάγη είναι μια συμφωνία προκειμένου να ληφθούν τα μέτρα που θα οδηγήσουν σε μία αύξηση κατά περισσότερο από 2 βαθμούς Κελσίου της θερμοκρασίας στον κόσμο. Και επίσης να έχουμε μία συμφωνία η οποία θα μπορεί να προσαρμοστεί στο μέλλον με βάση τα επιστημονικά δεδομένα. Το πρόβλημα με όλες αυτές τις διαπραγματεύσεις και τις διασκέψεις είναι ότι όλοι έχουν πολύ αυστηρή εντολή και όλοι οι υπουργοί παίρνουν τηλέφωνο την πρωτεύουσα και ρωτάνε τι περιθώρια ελιγμών έχουν. Έχουμε όμως να κάνουμε με μεγάλες οικονομικές δεσμεύσεις εδώ, μεγάλες μεταφορές κονδυλίων προς τις αναπτυσσόμενες χώρες και μεγάλες συνέπειες για τη βιομηχανία μας. Οπότε, πολύ απλά, από κάποια στιγμή και πέρα, οι Υπουργοί Περιβάλλοντος δεν είναι αρκετά υψηλά στην ιεραρχία για να λάβουν τέτοιου είδους αποφάσεις. Χρειάζονται ηγέτες κρατών και κυβερνήσεων για να λάβουν τόσο φιλόδοξες αποφάσεις ή αν όχι οι ηγέτες των κρατών, τουλάχιστον οι Υπουργοί Οικονομικών. Ο Βρετανός Πρωθυπουργό έχει καταστήσει σαφές τα τελευταία, τις τελευταίες ημέρες ότι θα παραστεί στην Κοπεχάγη. Οπότε αυτό που πρέπει να πάρουμε από την Επιτροπή μας και αυτό που πρέπει να ρωτήσουμε τις κυβερνήσεις μας είναι αν οι Υπουργοί Οικονομικών και αν οι Πρωθυπουργοί μας είναι διατεθειμένοι να πάνε στην Κοπενχάγη και να λάβουν αυτές τις σημαντικές αποφάσεις. Διαφορετικά θα μας απογοητεύσουν όλους. Ευχαριστώ τον κύριο Ντέιβις, ο κύριος Λίζε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, γιατί αυτό το θέμα είναι μοναδικό, γιατί δεν μπορούμε να το συγκρίνουμε με άλλα πολιτικά θέματα. Στα άλλα πολιτικά θέματα πάντα μπορούμε να καταλήγουμε σε συμβαστικές λύσεις, ενώ εδώ τα πράγματα δεν είναι έτσι. Ο πρόεδρος Σαρκοζή πέρσι είχε κάνει μια ομιλία για τα κλιματικά θέματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είπε ότι είναι σημαντικό γιατί είναι καλύτερα τα πράγματα γιατί πράγματι έχουμε επιστημονική εμπειρογνωμοσύνη και είναι απαραίτητο τα επόμενα 10 χρόνια να μειώσουμε τι εκπομπέ των αερίων θερμοκήπιων, αλλιώ οι επερχόμενε γενιές θα έχουν τεράστια προβλήματα να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση. Λοιπόν, πλησιάζουμε σε ένα σημείο καμπή. πρέπει να κάνουμε τι απαραίτητε ενέργειε για να μην είναι ασήκωτο το βάρο για τι επόμενε γενιές. Πρέπει να το λάβουμε λοιπόν αυτό σοβαρά. Ε, μου είπε ένα εμπειρογνώμων ότι αν γίνει ένα ατύχημα, ένα, ένα, ένα βάγιο πέντε χιλιόμετρα από τι ακτέ, δεν μπορεί κανεί να έχει μια εμπειρογνωμοσύνη που λέει ότι μπορεί να κολυμπήσει κανεί 4 χιλιόμετρα. Αλλά αυτό δεν λύνει το πρόβλημα. Επομένω, είναι απαραίτητο εμεί να κάνουμε τι απαραίτητε προσπάθειε που θα φτάσουν μέχρι εκεί που χρειάζεται. Είναι ένα δύσκολο λοιπόν θέμα. Εγώ από αυτά που ακούω στι ΗΠΑ δεν μπορώ να είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξο. Κάτι πιο συγκεκριμένο. Εγώ υπήρξα η εισηγητή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη συμπερίληψη των εναρίων μεταφορών στην εμπορία εκπομπών και αυτό πρέπει να είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα στην Κοπενχάγη. Εμεί έχουμε μια ευρωπαϊκή λύση, αλλά αυτή η ευρωπαϊκή λύση δεν θα μπορέσει να λύσει τα παγκόσμια προβλήματα ε, σε επίπεδο παγκόσμιο. Εμείς βλέπουμε να υπάρχει μία, ένας διπλασιασμός των εκπομπών από το 1990 στην εναέρια κυκλοφορία και επομένως είναι απαραίτητο εμείς να συμπεριλάβουμε αυτή την προβληματική στην Κοπενχάγη για τις εναέριες μεταφορές και θα πρέπει εκεί να θέσουμε κάποιους φιλόδοξους στόχους σαν Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης θα πρέπει να κάνουμε σαφές προς τις αναπτυσσόμενες χώρες της διαπραγματεύσεις μας ότι μία πτήση από την Κίνα ως το Λονδίνο ή από την Ινδία ως τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί σαν στοιχείο των στόχων των αναπτυσσόμενων χωρών. Τα άτομα αυτά τα οποία πετούν από τις χώρες αυτές τις Πολιτείες ή στην το Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι αυτοί οι οποίοι πλήττονται από την κλιματική αλλαγή, είναι αυτοί οι οποίοι έχουν λεφτά να πληρώσουν μια τέτοια πτήση και επομένω δεν πρέπει να του αντιμετωπίσουμε σαν να είναι απλώ πολίτε αναπτυσσομένων χωρών. Ένα άλλο θέμα είναι οι θαλάσσιε κυκλοφο... και υπάρχει μια πολύ μεγάλη δυνατότητα μέσα στα πλαίσια του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού να υπάρξει μια κοινή προσπάθεια για τη μείωση αυτού του, αυτών των εκπομπών Επίσης, εγώ είμαι απόλυτα απογοητευμένος για το γεγονός ότι οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων στο Pittsburgh δεν αναφέρθηκαν καθόλου στα ζητήματα αυτά. Τέλος, τελευταίο θέμα. Η χρηματοδότηση. Εγώ καταλαβαίνω όλα αυτά. Καταλαβαίνω όλους αυτούς που λένε ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες θα πρέπει να δώσουν χρηματοδότηση για τη μεταλαμπάδευση τεχνολογίας και την προστασία του κλίματος και την ε, προσαρμογή των αναπτυσσομένων χωρών στην κλιματική προστασία. Δεν πρέπει εμεί όμω να κάνουμε το λάθο να πιστεύουμε ότι αυτή η μεταφορά χρημάτων και τεχνολογία είναι το κύριο ζήτημα. Το κύριο ζήτημα που μα απασχολεί πρέπει να είναι η αντιμετώπιση τη κλιματική αλλαγή. και εμεί πρέπει να παίξουμε ένα ρόλο ηγέτη εναντί των αναπτυσσομένων χωρών και να πούμε ότι αν <clears throat> η κλιματική αλλαγή πάρει τη μορφή που αναφέρουν οι εμπειρογνώμονες, τότε αυτοί που ζουν στι αναπτυσσόμενες χώρε θα πληγούν πολύ περισσότερο από αυτούς που ζουν στις αναπτυγμένε χώρε. Δεν είναι μονάχα θέμα ότι δίνουμε 2 δισεκατομμύρια και αν δεν δώσουμε αυτά τα 2 δισεκατομμύρια απλώ δεν είχαμε μια συμφωνία. Θα πρέπει να αναλάβουμε μια πραγματική ευθύνη, να είμαστε ηγέτες αυτού του αγώνα για την προστασία από την κλιματική αλλαγή στι αναπτυσσόμενε χώρε. Και προσυπογράφω αυτά που είπε και ο Καρλ Χάιντ Φλόρεν για τη σωστή χρησιμοποίηση αυτών των ποσών που θα δώσουμε στι αναπτυσσόμενε χώρε και τον, την εποπτεία τη σωστή του χρηματοδότηση. <clears throat> Είναι απαραίτητο λοιπόν να τονίσω ότι αυτά τα οποία προτείνει η Κομισιόν προς το παρόν δεν είναι αρκετά. Υπάρχουν κάποια ρεφλέξ, υπάρχει μια ε, σταθερή στάση στα κράτη-μέλη για την ε, ανάγκη να εμπλέξουμε και τις Ηνωμένε Πολιτείες, εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ω κοινοβούλιο να έχουμε έλεγχο στα κονδύλια αυτά. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα ταμείο το οποίο είναι καθαρά διακυβερνητικού χαρακτήρα, το οποίο δεν ελέγχεται καθόλου από πολιτικού όπω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό πρέπει να το εξηγήσουμε στου πολίτε μα. Θα πρέπει να τονίσουμε στην Κομισιόν ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει ένα στοιχείο στον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο όμω να είναι ελέγξιμο από του κοινοβουλευτικού και να μπορούμε να το αιτιολογήσουμε στου πολίτε μα. Το θέμα τη εμπορία εκπομπών. Εγώ συμφωνώ με τον Καρλ Χάτ Φλόρεν. Δεν μπορούμε να παραμείνουμε μοναχά στο θέμα τη εμπορία εκπομπών, ούτε καν σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση. Πάνω από 50% των εκπομπών στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα <clears throat> προέλθουν από τομεί οι οποίοι δεν καλύπτονται καν από την από την εμπορία εκπομπών. Γιατί η χαλιβουργία και η παραγωγή τσιμέντου να είναι υπεύθυνε για τις εκπομπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επομένως να πληγούν από τις συμφωνίες που θα κάνουν σε διεθνές επίπεδο. Θα πρέπει όλοι οι εμπλεκόμενοι τομείς <clears throat> να συμπεριληφθούν στην πρόταση της Κομισιόν και υπάρχει η πρόταση της Νορβηγίας η οποία ζητά ένα μέρος χρηματοδότησης να γίνεται από τα κράτη και όχι μονάχα από τις επιχειρήσεις και αυτό το βρίσκω κάτι θετικό και για τη διατήρηση ανταγωνιστικότητας. Τέταρτο, τελευταίο, ζητούμε μια πολιτική ηγεσία. Και έχει απόλυτο δίκιο ο Κρις Davis. Θα πρέπει να τραβήξουμε τα αυτιά και των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων και να τους πιέσουμε να αναλάβουν αυτήν την ευθύνη αλλά επίσης θα πρέπει να πιέσουμε και τον κύριο Ομπάμα, ο οποίος έχει κάνει λαμπρές και μεγαλεπίβολες δηλώσεις, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι το οποίο είναι απαραίτητα, απαραίτητο να γίνει είπε ότι θα πάει στην Κοπενχάγη ο κύριος Ομπάμα, αλλά δυστυχώ όχι για την κλιματική, τη συνδυάση κλιματικής αλλαγής, αλλά για να υποστηρίξει την πρόταση του Σικάγου να είναι οικοδεσπότη των μελλοντικών Ολυμπιακών Αγώνων του 2016. Αυτό λοιπόν δεν είναι κάτι που μπορούμε να υποστηρίξουμε. Η κυρία Ζορντάν Σίζελ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρα. Θα ήθελα να συμφωνήσω με τους συναδέλφους που τόνισαν ότι θα πρέπει να περιμένουμε συγκεκριμένες προτάσεις από τους ηγέτες της Ιφιλίου στην Κοπενχάγη και εφικτές προτάσεις. Εδώ θα ήθελα να αναφερθώ σε μια άλλη χώρα πέραν της Κίνας, την Ινδία. Θεωρώ ότι η προσέγγιση τους απέναντι στην κλιματική αλλαγή είναι ιδιαίτερα ανησυχητική. Επίσης, έχουμε πολλές ανησυχίες και όσον αφορά τη στάση του Προέδρου Ομπάμα και τον ΙΠΑ. Κάτι άλλο τώρα όμως. Η κλιματική αλλαγή είναι οριζόντιο φαινόμενο. Αρχικά συζητούσαμε το θέμα της κλιματικής αλλαγής μόνο στα πλαίσια της προστασίας του περιβάλλοντος. Τώρα όμως τα πράγματα έχουν αλλάξει και το συζητάμε οριζοντίως το θέμα. Πέρα από εμάς, μία ακόμη επιτροπή που ασχολείται με το θέμα είναι η Επιτροπή Βιομηχανίας, η Ήτρε. Και χτες συζητούσαμε αυτό το ψήφισμα περισσότερο από τρεις ώρες καταλήξαμε ότι είναι ένα καλή βάση, αλλά υπάρχουν κάποιες ελλείψεις και γι' αυτό κάναμε κάποιες προτάσεις για τροποποίηση. Αυτό που θα ήθελα να ζητήσω από τα μέλη της Επιτροπής σας είναι να λάβετε υπόψη τις προτάσεις τροποποίησης της Επιτροπής Βιομηχανίας γιατί πρέπει να θυμάστε ότι έχουμε και εμείς πολλές αρμοδιότητες στον τομέα αυτό όπως για παράδειγμα ανάπτυξη τεχνολογιών με χαμηλή χρήση άνθρακα κάτι που μπορεί να γίνει εφικτό μόνο αν έχουμε καλή ανταλλαγή τεχνολογίας και συνεργασία έρευνας και επιχειρήσεων. Και επίσης εδώ πρέπει να δούμε και πώς θα εμπλέξουμε και τις αναπτυσσόμενες χώρες προκειμένου να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνδέσεις μεταξύ κρατών που θα επιτρέπουν και την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας. Κάτι άλλο που μας απασχολεί ιδιαίτερα είναι η, η μετεγκατάσταση των ε, εκπομπών. Θεωρώ ότι το να χρησιμοποιούμε κάτι τέτοιο είναι αρνητικό. Χρειαζόμαστε νέες τεχνολογίες που θα προλαμβάνει αυτή την κατάσταση. Πρέπει λοιπόν να γίνει έκκληση στις υπόλοιπες βιομηχανικές χώρες του κόσμου να ενώσουν τις δυνάμεις τους με την Ευρωπαϊκή Ένωση για να το επιτύχουμε αυτό. Και περνάω τώρα στις ανανεώσιμες ενέργειες και γενικά την ενέργεια. Πρέπει να τονίσουμε και την ανάγκη αύξησης της αποδοτικότητας της ενέργειας που χρησιμοποιούμε τώρα και την χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Και όσον αφορά τα ορεικτά καύσιμα που είναι πολύ σημαντικά για χώρες όπως η Κίνα και η Ρωσία, θα πρέπει και εδώ να επιτύχουμε και τη χρήση πιο καθαρών τεχνολογιών και τη μεγαλύτερη συνεργασία σε διεθνές επίπεδο. Τέλος, αυτό που θέλουμε είναι να δώσουμε όθηση στην έρευνα και την ανάπτυξη γιατί αν βρούμε νέα μοντέλα τότε θα μπορέσουμε να έχουμε πιο γρήγορη και πιο αποτελεσματική ανταλλαγή τεχνογνωσίας με τον αναπτυσσόμενο κόσμο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ιλπαριού. Σας ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Επιτρέψτε μου πέραν της ικανοποίησης που μπορεί να αισθάνομαι δεδομένων των ισχυρών αυτών κατευθύνσεων και προσανατολισμών που αναφέρατε στο συγκεκριμένο σχέδιο ε, θέλω τώρα να αναφερθώ στη χρηματοδότηση και νομίζω ότι πρέπει να προχωρήσουμε περισσότερο στι οικονομικέ υποχρεώσει ε, και για να μπορέσουμε να πετύχουμε του στόχου μα και ταυτόχρονα να κάνουμε και αυτά τα οποία αναφέρουμε στο σχέδιο ψηφίσματο. Δηλαδή ότι ε, η Κοπεχάγη να παράσει τα αναγκαία κίνητρα για μια πράσινη νέα συμφωνία που θα δώσει όφηση στην οικονομική ανάπτυξη. Άρα πιστεύω ότι το σχέδιο ψηφίσματο θα πρέπει να αναφερθεί και στο ε, φόρο άνθρακα στα σύνορα. Ξέρουμε ε, τι γίνεται και την ανάγκη που υπάρχει μείωσης ε, με βάση τις διαπραγματεύσεις που γίνονται. πιστεύω λοιπόν ότι το, το πακέτο ενέργεια και κλίμα θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να δώσουμε περισσότερα κίνητρα στις ανεψόμενες χώρες για να ταυτούν συμφωνία. Νομίζω λοιπόν και έθεσα και γραπτό ερώτημα προς την Επιτροπή που πιστεύει ότι πρέπει να περιμένουμε την Κοπεχάγη και στη συνέχεια να έχουμε μία ε, έκθεση ε, και μία ανάλυση. Εγώ νομίζω από τώρα θα πρέπει να αναφέρουμε αυτό το οποίο εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυμούμε να πράξουμε ε, όσον αφορά αυτές τις διαρροές άνθρακα και να αναφέρουμε στο σχέδιο ψηφίσματος τους στόχους μας που θα μπορούσαμε για παράδειγμα να συμπεριλάβουμε εκεί που αναφέρουμε στις ε, ποσοστώσεις ε, ε, δωρεάν και το σύστημα ανταλλαγής εκπομπών να αναφέρουμε και τα, και κατάλληλα μέτρα τα οποία αφορούν την, την ηλεκτρική διασύνδεση, τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις. Νομίζω λοιπόν ότι θα μπορούσαμε να λάβουμε όλα αυτά τα στοιχεία υπόψη για να αναφέρουμε ακριβώς εν ώψη της Συνόδου Κορυφής Κοπενχάγης αυτό το οποίο θα ε, ε, πρέπει να κάνουμε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για την ε, συνοπτική σας παρουσίαση και για την ε, ε, βραχύτητα των λόγων σας. Θα δώσουμε το λόγο στην κυρία Κορτίνες. Σας ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Θα ήθελα να μιλήσω για το σημείο 17 Έρχομαι από την Αργεντινή, από τη Σύνοδο Κορυφή για την Αποψήλωση. Και το ψήφισμα των κοινοβουλίων εκεί ήταν ακριβώ αυτό. Ότι ε, η απερίμωση να συμπεριληφθεί συγκεκριμένα στην Κοπεχάγη. Θα προτείνω λοιπόν δύο ή τρει τροπολογίε που, που θα αναφερθούν στο εξή. Στο 17, εκεί όπου αναφέρεται η μείωση των εκπομπών από την αποψήλωση και υποβάθμιση των δασών και την υποβάθμιση του εδάφους να, και να αναφέρουμε και την απερίμωση. Επίσης, την ίδια παράγραφο. Μια άλλη ιδέα που είναι θεμελιώδης κατά την άποψή μου είναι η εξή. Η κοινή αγροτική πολιτική θα πρέπει να είναι συνεπής και συνεκτική με ε, ε, την κλιματική αλλαγή. Γιατί στι χώρε του Νότου τι γίνεται. Πληρώνει η Επιτροπή για να, για να κρυζώνουμε δέντρα, αμπελώνε, ε, ελαιώνες, ελαιόδεντρα. Αυτό όμω σημαίνει υποβάθμιση του εδάφου ε, και απορρίμωση. Ένα πράγμα είναι περιορισμός τη παραγωγή και ένα άλλο πράγμα να ξεριζώνουμε δέντρα. Είναι ε, ε, ε παράλογο και θα πρέπει να δούμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι ποιο σημείο μπορούμε να έχουμε τι πολιτικέ. Θα ήθελα και, και άλλε πολιτικέ ομάδε να με υποστηρίξουν αυτήν την τροπολογία. Πρώτα πρέπει να με συνεπεί με τον ίδιο μα τον εαυτό. Ε, ε, να κάνουμε τουλάχιστον ε, τι δικέ μα τι δουλειέ, το δικό μα το σπίτι και μετά να κοιτάμε τι κάνουν οι άλλοι. Και επίση στι γεωργικέ πολιτικέ ε, να συμπεριλάβουμε την ανάκτηση των δασών, την αναδάσωση. Γιατί καίγονται τα δάση, καταστρέφονται τα δάση. Πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Και κάτι άλλο στη χρηματοδότηση. Και το ζητούν και τρίτε χώρε. Να κάνουμε μια σαφή χειρονομία. Δηλαδή ότι σε αυτή τη δικασία προσαρμογή θα υπάρξουν ευρωπαϊκό κονδύλια η μνήμη του, η ιστορική του μνήμη είναι σαφή. Η Ινδία είπε κυριολεκτικά ότι εμεί πάμε ξυπόλοιποι. Και ε, τι έχουμε, έχουμε ε, το πολύ ένα μηχανάκι ή ένα, ή ένα ποδήλατο. Ε, καταλαβαίνετε. Ε, η Ινδία λοιπόν δεν έχει καμία σχέση με την Κοπεχάγη. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστέ. Άρα ένα, ένα που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε είναι ότι η Ευρώπη πρέπει να πληρώσει και να διορθώσει αυτά που έκανε μέχρι στιγμής με συγκεκριμένη χειρονομία, λαμβάνοντα υπόψη ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο πρόβλημα φτώχεια, αλλά σε πολλές περιπτώσεις capacity building, δηλαδή ε, δική τους ε, εσωτερική ικανότητα. Ε, και να σα πω και κάτι άλλο, ότι θα πρέπει να εισάγουμε μία σαφή ιδέα για το μετά την Κοπεχάγια. Όπω ακριβώ ήταν σαφέ, ήταν εύκολο να βάλουμε κριτήρια για τη μείωση των εκπομπών για τη βιομηχανία. Κοιτάξτε, να κάνουμε μαθηματικά μοντέλα που θα εφαρμόζει η βιομηχανία δεν υπάρχει πρόβλημα αλλά ε, σε, ε, στο καινούριο, ε, στην καινούργια θητεία πρέπει να ξέρουμε επί επιτόπου κάθε περιοχή, κάθε περιφέρεια, τι εκπέμπει, τι δάση, ε, ε είναι, ποιο έδαφο ε, θα απορροφά το, το διοξείδιο του άνθρακο και με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε ολοκληρωμένη πολιτική σε κάθε περιοχή. Η επιστήμη έχει προοδεύσει αρκετά και μπορούμε να εργαστούμε με συγκεκριμένα στοιχεία. Μέχρι στιγμή δεν είχαμε στοιχεία. Να μιλάμε λοιπόν μόνο για τη βιομηχανία νομίζω ότι είναι ε, να ασχολούμαστε με ένα πολύ μικρό ποσοστό του θέματος. Αν θέλουμε να το καλύψουμε σφαιρικά, με συστηματικό τρόπο και να δεχτούμε ότι το, θέμα είναι περίπλοκο, να συμπεριλάβουμε τις επιτόπου περιφέρειες και την ανάλυση τους. Πρόταση. Με συγκεκριμένε ημερομηνίε και με συγκεκριμένα στοιχεία για να εργαστούμε για το θέμα των εκπομπών επιτόπου στην κάθε περιοχή ξεχωριστά. Ευχαριστώ. Äh, Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι αυτό το οποίο συζητούμε σήμερα είναι ένα έγγραφο το οποίο είναι σημαντικό. Η διάσκεψη Κοπενχάγης όμως θα έχει τουλάχιστον δύο διαστάσεις, μία επιστημονική και μία πολιτική. Η πεποίθησή μου είναι ότι η πολιτική διάσταση θα είναι η πιο σημαντική. Τι σημαίνει αυτό. Ένα παγκόσμιο πρόβλημα δεν μπορεί να επιληθεί με τοπικά μέτρα. Η Ευρώπη μπορεί να δώσει ένα παράδειγμα, ένα θετικό παράδειγμα και όπως είπαμε και στο παρελθόν μπορεί να προχωρήσει και σε ένα επίπεδο συμμόρφωσης που δεν το επιτυγχάνουν τα άλλα κράτη. Αλλά δεν θα πετύχουμε τίποτα αν οι δύο μεγαλύτεροι ρηπαντέ, δηλαδή οι Ηνωμένε Πολιτείε και η Κίνα, δεν πιστούν να μειώσουν τι εκπομπέ τους. Ο κ. Κάρδιον, ο Υπουργό Περιβάλλοντος τη Σουηδία, είχε πει ότι μπορεί κανείς να περιμένει από τι Ηνωμένε Πολιτείε να πράξουν ό,τι το δυνατό. Αλλά ξέρουμε από την εποχή του πρωτοκόλλου του Κιώτο ότι το μεγαλύτερο που μπορεί να κάνουν, το πιο πολύ μπορεί να κάνουν οι Αμερικανοί, δεν είναι επαρκές. Πρέπει λοιπόν να είμαστε σαφείς απέναντί τους. Ο Ζισκάρ Ντεστέν, ο οποίος ήταν ο πρόεδρος της ε, συντακτικής συνέλευσης, όταν προετοιμάζαμε το Σύνταγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι αντίπαλος, αλλά εταίρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Προκύψει λοιπόν σημαντικές συνέπειες από όλα αυτά τα γεγονότα. <clears throat> Όταν τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν αντιπροσωπεύτηκαν σωστά από τους ηγέτες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρξει, όπως προτάθηκε από, το, από κάποιους ομιλητές, να υπάρξει επαφή και μέσω ίντερνετ των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πολιτών των Ηνωμένων Πολιτειών. Η άμεση δημοκρατία, η άμεση ηλεκτρονική δημοκρατία δεν λαμβάνεται υπόψη σοβαρά στην Ευρωπαϊκή Ένωση όταν υπάρχουν σημαντικά προβλήματα. Εμείς οι αντιφρονούντες πολλές φορές δεν μπορούμε να παρουσιάσουμε τις απόψεις μας. Αλλά στην Κοπεχάγη θα πρέπει να υπάρξει μια σωστή αντιπροσώπευση του πληθυσμού πολλών χωρών που δεν θα είναι παρούσες. Εγώ νομίζω ότι δεν είναι λογικό οι τέσσερις από τις πέντε παρεμβάσεις να αναφέρονται στις ευθύνε των ΗΠΑ αλλά δεν συνεχίζουν στο θέμα αυτό. Είμαι πεπισμένος ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρώπη θα πρέπει μέσα στα πλαίσια αυτής της κατάστασης να εκπροσωπήσει και τις 27 χώρες της και τα 750 εκατομμύρια πολιτών της. Αυτό όχι μονάχα προς το κοινό, το δημόσιο συμφέρον, αλλά και γιατί με τον τρόπο αυτό θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της η Ευρωπαϊκή Ένωση και να προχωρήσει να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την περιστολή αυτών των εκπομπών. Ίσως λοιπόν δεν εναπόκειται σαν μένα ως ανεξάρτητο βουλευτή να κάνω προτάσεις. Αλλά αν θέλουμε να δείξουμε ότι είμαστε υπεύθυνοι, γιατί αυτή η ευθύνη να μην περιλαμβάνεται στο ψηφισμά μας και γιατί να μην στείλουμε εκπροσώπους στην Κοπεχάγη από την χωρία αυτών που θέλουν πράγματι να γίνει κάτι για τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κυλακάκης έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ξεκινήσω με την εξής παρατήρηση. Μιλάμε πολύ για τη χρηματοδότηση, αλλά δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι στον τελευταίο χρόνο ξοδεύτηκαν περίπου 2-3 εκατομμύρια ευρώ από τις, αναπτυσσο... από αναπτυγμένες χώρες για την αντιμετώπιση οικονομικής κρίσης. Αυτό σημαίνει ότι όταν υπάρχει πολιτική βούληση μπορούν να βρεθούν χρήματα, αν και στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν χρήματα από το μέλλον, κυρίως με δανεισμό. Μια δεύτερη παρατήρηση είναι πώς θα χρησιμοποιήσουμε και πόσο δημόσιους πόρους θα πρέπει να θυμόμαστε ότι η βασική αρχή οριπένων πληρώνει ισχύει τουλάχιστον για τη μελλοντική ρήπανση και εδώ και θα πρέπει να τη λαμβάνουμε υπόψη σε σχέση με τη δημόσια χρηματοδότηση. Όπου είναι εφικτό και δίκαιο πρέπει η αρχή οριπένων πληρώνει να εφαρμόζεται και εδώ. Τώρα έρχομαι στο κεφάλαιο ε, για τις αεροπορικές μεταφορές και την αυτιλία που ε, θεωρώ ότι έχει ιδιαίτερη σημασία σε αυτό το ψήφισμα. Καταρχήν βάζουμε δύο, τους δύο αυτούς κλάδους μαζί. Πρέπει να γνωρίζουμε όμως ότι είναι ουσιαστικά διαφορετική κλάδη από πλευράς ρήπανσης. Οι αερομεταφορές ρηπαίνουν πολύ περισσότερο από ότι η ναυτιλία που είναι ο ενεργειακά αποδοτικότερος τρόπος μεταφορών προσωπικά πιστεύω ότι και οι δύο κλάδοι πρέπει να περιληφθούν στη συνολική προσπάθεια. οι στόχοι όμως που θα πρέπει να τεθούν πρέπει να λάβουν υπόψη την ενεργειακή αποδοτικότητα και τους στόχους τους οι οποίοι τίθενται για τις χερσαίες μεταφορές οι οποίοι φοβούμε είναι πολύ λίγο φιλόδοξοι. οι χερσαίες μεταφορές εντός της ευρωπαϊκής ένωσης έχουν τη συντριπτική, τη μεγάλη πλειοψηφία της ρήπανσης του συνολικού κλάδου μεταφορών. Τα αυτοκίνητα μόνο αναλογούν στη μισή από τη ρήπανση. Δεν μπορεί λοιπόν οι δύο κλάδοι που ανταγωνίζονται τις χερσαίες μεταφορές να έχουν τελείως διαφορετική μεταχείριση από πλευράς στοχοθεσίας, από πλευράς targeting. Και μάλιστα ο περισσότερο σχετικά ρηπογόνος, οι χερσαίες μεταφορές να έχουν διακριτική μεταχείριση. Επίσης, σε σχέση με την ε, παράγραφο 19, νομίζω ότι δεν είναι σωστό να προεξοφλήσουμε την αποτυχία των διαπραγματεύσεων στον IMO και τον ICAO. Πρέπει να στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα, χωρίς όμως να προεξοφλούμε την αποτυχία. Με τα δεδομένα αυτά ε, ε, θα καταθέσω δύο τροπολογίες. Μία τροπολογία στην παράγραφο 18, ε, θα διαβάσω το αγγλικό κείμενο γιατί αυτό έχω, ε, ε, εκεί που λέει «Insist that the international aviation and maritime sectors should be subject to the same target as other industries», μία παρένθεση η οποία θα λέει «including land transport», έτσι ώστε να συνδέονται αυτοί οι τρεις ανταγωνιστικοί μεταξύ τους κλάδοι και στην παράγραφο 19 εκεί που λέει urges the EU with a view to the failure of the ε, ICAO and IMO talks να αντικατασταθεί το with a view to the failure με το in case of a failure. Δεν μπορούμε να προεξοφλήσουμε ότι θα αποτύχουν, πρέπει να πάρουμε μέτρα, αλλά ο στόχος καταρχήν θα πρέπει να είναι να πετύχουν αυτές οι διαπραγματεύσεις. Αυτός είναι και ο στόχος του Συμβουλίου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ο Μπάσα Ικούτ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι πολλοί από τους ομιλητές αναφέρθηκαν στο στόχο της μη αύξησης πέραν των δύο βαθμών που είναι ένας κεντρικός στόχος μας. Αλλά πρέπει να πω ότι αυτός ο στόχος δεν είναι στόχος μονάχα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή τη στιγμή. Είναι ένας στόχος τον οποίο τον έχουν υποστηρίξει στη συνεδρίαση των G20. Εγώ έρχομαι από τον επιστημονικό κόσμο και εργάζομαι για το θέμα αυτό εδώ και πάρα πολύ καιρό. Για να πετύχουμε αυτό το στόχο του να μην ξεπεράσουμε τους δύο βαθμούς, θα πρέπει να φτάσουμε σε μείωση των εκπομπών κατά 40% για να έχουμε πιθανότητα 50% να πετύχουμε το στόχο αυτό του 2%. Λοιπόν, για να τηρήσουμε αυτό το στόχο πρέπει να έχουμε τις κατάλληλες πολιτικές. Για την κυρία Γκροστέθ η οποία πρέπει να, είμαστε, πρέπει να είμαστε αξιόπιστοι προς τα έξω. Κοιτάξτε την Κίνα η Κίνα αυτή τη στιγμή δημιουργεί αιωλικέ εγκαταστάσει. Σε δύο χρόνια θα έχουν τη μεγαλύτερη παραγωγή αιωλική ενέργεια στον κόσμο. Αυτό κάνει η Κίνα σήμερα. <clears throat> Αυτό συμβαίνει όταν υπάρχει πολιτική θέληση. Μπορεί να υπάρξει μια αλλαγή. Μπορούμε να κινηθούμε προ μια πράσινη οικονομία. Αυτό πρέπει να πράξουμε. Γι' αυτό ζητώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι πιο σαφή σε σχέση με τον στόχο του των δύο βαθμών και να κάνει τα απαραίτητα μέτρα για να φτάσει στο στόχο αυτό, να έχει αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα στη χρήση ενέργειας, αύξηση των ανανεωσίμων ενεργειών, να μην μιλάμε μόνο για τη μείωση των εκπομπών ρήπων, αλλά να δούμε και ποια είναι η δυνατότητα που μπορεί να αποκομίσει η ευρωπαϊκή βιομηχανία. Αυτό θα μας κάνει αξιόπιστος εναντί των Κινέζων και των Αμερικανών. Η Κίνα γίνεται πια ο μεγαλύτερος παραγωγός ενέργειας σε όλους τους τομείς ακόμα και στην παραγωγή ενέργειας από άνθρακα. Αλλά και στην ηλιακή ενέργεια, λέει ο κύριο Σέικουτ. Μην δείτε μονάχα τη μία πλευρά, δείτε και την άλλη πλευρά. Η Κάτριν Φαν Μπρέμπτ έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, θα είμαι πολύ σύντομη γιατί ήδη ακούσαμε εξαιρετικές παρεμβάσεις. Νομίζω ότι είναι εξαιρετικό σημείο εκκίνησης ε, το κείμενο που έχουμε και είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει μεγάλη συνένεση στα πλαίσια του Κοινοβουλίου πρέπει βεβαίως να ενισχύσουμε αυτό το κείμενο. Εγώ αυτό που θέλω είναι όντως να έχουμε συγκεκριμένους στόχους, αλλά το εξίσου σημαντικό είναι να επιτύχουμε αυτούς τους στόχους. Αυτή τη στιγμή στρεφόμαστε στις αναπτυσσόμενες χώρες, αλλά παράλληλα δεχόμαστε, πρέπει να δεχτούμε και φιλόδοξους στόχους για εμάς τους ίδιους. Εκεί είναι που βλέπω κάποιες αδυναμίες στο κείμενο, γιατί πρέπει να είμαστε πολύ αξιόπιστοι και πρέπει λοιπόν να μιλήσουμε για συγκεκριμένες γραμμές του προϋπολογισμού που θα αξιοποιήσουμε για να επιτύχουμε τους στόχους μας. Έχουμε να κάνουμε με ένα ακόμη θέμα το οποίο αποτελεί σημαντική πρόκληση. Τις αναθεώσιμες πηγές ενέργειας. Μέχρι στιγμής έχουμε κάνει λίγα στον τομέα αυτό. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να αξιοποιήσουμε και το ψήφισμα για να τονίσουμε τη σημασία των αναπτυσσόμενων πηγών ενέργειας. Θεωρώ ότι και την αιωλική ενέργεια και την ηλιακή πρέπει να τις αξιοποιήσουμε ιδιαίτερα. Ειδικά όσον αφορά την αιωλική ενέργεια στο βορρά έχουμε πολλές δυνατότητες. Πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει κίνητρα στα κράτη-μέλη να ασχοληθούν με το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ο Ματίας Γκρότε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εδώ ελέγχθη ότι οι στόχοι δεν πρέπει να τεθούν τόσο εκπεφρασμένα γιατί ενδεχομένως δεν θα είμαστε σε θέμα δεν θα είμαστε σε, δυνατό, δεν θα είμαστε σε θέση να τους πετύχουμε. Εδώ έχουμε να αντιμετωπίσουμε θέματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά όπως αναφέρεται και στο ψήφισμά μας την, την ε, οικονομική κρίση παράλληλα με την, με την κρίση του, του περιβάλλοντος. Πρέπει όμως να συνδέσουμε αυτά τα δύο στοιχεία. Νομίζω ότι είναι απαραίτητο να εξασφαλίσουμε ότι θα έχουμε φιλόδοξους στόχους και ότι θα έχουμε και τα εργαλεία με τα οποία θα μπορέσουμε να πετύχουμε αυτούς τους στόχους. Και για μένα το πιο σημαντικό στοιχείο είναι η μεταλαμπάδευση της τεχνολογίας. Αυτή τη στιγμή έχουμε φωτοβολταϊκά συστήματα τα οποία παραδίδονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από άλλες περιοχές του κόσμου και τα οποία δεν λειτουργούν και κάποια στιγμή δεν έχουν κανένα αποτέλεσμα. Εμείς όμως ως Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι δίνουμε την κατάλληλη τεχνολογία στις άλλες χώρες και αυτά τα οποία δίνουμε παραγματικά χάρη στην Κίνα να είναι επαρκούς τεχνολογίας και να μην βλέπουμε τα πράγματα μονάχα μέσα από ροδόχρωα γυαλιά. Θα πρέπει επίσης να δούμε τι γίνεται και με τις αιωλικές τουρμπίνες. Αυτή τη στιγμή έχουμε χρόνο παράδοσης 3 με 4 χρόνια και δεν υπάρχει η, η ικανότητα ανάπτυξης αυτής της τεχνολογίας πολλές φορές λόγω έλλειψης χρηματοδότησης. Το σημείο 18 και 19, αυτά που είπε ο κύριος Λίζε για τις θαλάσσιες και εναέριες μεταφορές. Πρέπει πράγματι τα θέματα αυτά να αντιμετωπιστούν στην Κοπενχάγη. Ο ΙΚΑ, ο Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας, έχει ζητήσει έχει συζητήσει ήδη το θέμα αυτό. Εμείς νομίζω ότι έχουμε πραγματικά σωστά επιχειρήματα να συμπεριληφθεί το θέμα αυτό στην ε, συζήτηση Κοπενχάγης. Εμείς έχουμε πάντα αναφέρει τις αποφάσεις του ΙΚΑΟ, αλλά δεν πρέπει να παραμείνουμε μονάχα σε ένα φραστικό επίπεδο. Θα πρέπει η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κοπεχάγη να τονίσει ότι πρέπει το θέμα αυτό να αντιμετωπιστεί και αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί μονάχα με παγκόσμια φράση, υπάρχει ένα σύνδεγμα, σύστημα το οποίο λειτουργεί, που είναι η εμπορία εκπομπών. Μπορούμε να μιλήσουμε και για φορολογικά κίνητρα ή αντικίνητρα, αλλά είναι απαραίτητο η Ευρωπαϊκή Ένωση να ξέρει ότι αν δεν μπορεί να εναρμονίσει τη φορολογία στο εσωτερικό της, δεν μπορεί να την επιτύχει σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι απαραίτητο λοιπόν εμεί να βάλουμε το πρώτο λιθαράκι και να παροτρύνουμε και του άλλου εταίρου μα στις διαπραγματεύσει να προχωρήσουν προ την κατεύθυνση αυτή, δηλαδή να συμπεριληφθεί και το θέμα της θαλάσσιας, των θαλάσσιων μεταφορών και των εναέριων μεταφορών στην συνολική προβληματική. Ζέμπα. Ευχαριστώ κύριε Πρόβλε. Κυρίε και κύριοι, θέλω να σα υπενθυμίσω ότι εμεί ω πολιτικοί θα πρέπει να βασίζουμε την ε, απόφασή μας στην εμπειρογνωμοσύνη των επιστημόνων αλλά και πάνω στην απλή ανθρώπινη κοινή λογική. Πριν από 100 χρόνια ξεκίνησε η θεωρία της σχετικότητος, η θεωρία τη κβαντική με τον Πλάνκ και άλλους. Όλα αυτά ήταν σημαντικά στοιχεία της ε, γνώσης στον κόσμο μας, αλλά το σημαντικό ήταν να μπορέσουν αυτές οι γνώσεις οι οποίες ξεκίνησαν στο επίπεδο μιας μικρής ομάδας επιστημόνων να γίνουν κτήμα όλων των πολιτών στις χώρες μας. Αν δούμε λοιπόν το θέμα της κλιματικής αλλαγής. Μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι υπάρχει αυτό το φαινόμενο. Αυτό είναι γενικά αποδεκτό. Η μεγάλη πλειοψηφία των επιστημόνων το αποδέχονται. Το δεύτερο πρόβλημα όμως, και εδώ θέλω να εστιάσω, είναι ότι αυτό θα πρέπει να γίνει κατανοητό και σε όλους τους πολίτες υπάρχει πάντα μια κοινότητα αντιφρονούντων οι οποίοι λένε ότι ένα πολύπλοκο σύστημα όπως ένα, το σύστημα της, ε, του κλίματος στην ε, γη μας δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να αντιμετωπιστεί με αλλαγές μονάχα σε μία, σε μία ισορροή όπως είναι αυτή των εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακος και ότι τα μοντέλα με υπολογιστές πολλές φορές είναι υπερβολικά πολύπλοκα και δεν δίνουν ε, μονοσήμαντες αποφάσεις. Ε, απαντήσεις. Πρέπει λοιπόν εμείς να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση και στην οικονομική μας πολιτική για να επηρεάσουμε την κλιματική αλλαγή. Επομένως, νομίζω ότι είναι απαραίτητο από τη δική μας πλευρά να έχουμε και μεγαλύτερη προσοχή στις προϋποθέσεις για να μπορέσει η Ευρώπη να αναλάβει ευθύνες στον τομέα της κλιματικής αλλαγής. Νομίζω για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό να εξασφαλίσουμε και το ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία δεν θα πληγεί μονομερός από όλες αυτές τις ενέργειες. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε λοιπόν ότι υπάρχει ισότηση συνδικών ανταγωνισμού για την ευρωπαϊκή βιομηχανία σε παγκόσμιο επίπεδο. και είναι ένα πολύμορφο και πολυεδρικό φαινόμενο το φαινόμενο της, κλασική, της ε, κλιματικής αναλλαγής και δεν μπορούμε να το δούμε μονάχα από μία σκοπιά όπως αυτή που παρουσιάζεται από πολλούς επιστήμονες. Επίσης στον τομέα της ενεργειακής αποδοτικότητας νομίζω και εδώ στην Ευρώπη έχουμε μεγάλη δυνατότητα να επιτύχουμε ε, σημαντικές πρόοδους γιατί οι τεχνολογίες που έχουμε μπορούν να είναι επιτυχείς σε παγκοσμίο επίπεδο. Εδώ θα μπορούσαμε μαζί με τους εταίρους μας να αναλάβουμε την ευθύνη κοινή δράση. Επίσης όμως θα πρέπει η Ευρώπη να είναι και πρωτοπόρο σε ό,τι αφορά την δημιουργία θέσεων απασχόληση στον τομέα αυτό. Τέλος το θέμα των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας. Είναι οι δύο μεγαλύτερη εκπομπή ε, διοξιδίου του άνθρακος και καλύπτουν σχεδόν το μισό των εκπομπών σε παγκοσμίο επίπεδο. Κατά την άποψή μου η Κίνα όμως έχει προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό σε ό,τι αφορά τη χρησιμοποίηση πράσινης ενέργειας και στις ε, συζητήσεις Κοπενχάγης δεν είναι η Κίνα που θα είναι το πρόβλημα. Είναι περισσότερο η Ινδία και άλλες χώρες BRIC οι οποίες θα είναι πρόβλημα μαζί με τις ε, Ηνωμένες Πολιτείες. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το πώς θα κινηθεί το Αμερικανικό Κογκρέσο έχει 18 εργάσιμες μέρες μονάχα το Κογκρέσο στο τέλος του χρόνου και η κυριαρχούσα συζήτηση αυτή τη στιγμή συζήτηση για τα θέματα υγειονομικής περίθαλψης. Και θα μετρηθεί η επιτυχία του Πρόεδρου Ομπάμα από το αν θα περάσει το θέμα της υγειονομικής περίθαλψης ή όχι στην πολιτική του. Δεν έχει λοιπόν το Κογκρέσο χρόνο να ασχοληθεί με την κλιματική αλλαγή. Είναι πάρα πολύ πιθανό ότι δεν θα υπάρξει καμία απόφαση σε επίπεδο Αμερικανικού Κογκρέσου και γι' αυτό εμείς θα πρέπει να προσορμόσουμε την, την ε, δική μας διαπραγματευτική τακτική. Εμείς λοιπόν δεν θα πρέπει να απογοητευτούμε από την Κοπενχάγη αν δεν υπάρξουν αποτελέσματα. Θα πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπαθίες μας λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι ΗΠΑ είναι πολλές φορές το μεγαλύτερο εμπόδιο. Εγώ περιμένω λοιπόν τώρα από τη νέα ε, Κομισιόν να μπορέσει να έχει μια καλύτερη αντιμετώπιση των επιπτώσεων που προέρχονται σε επίπεδο υδάτινων πόρων από την κλιματική αλλαγή σε ό,τι αφορά παραγωγός χάρη τις πλημμύρες, την αποτυχία των συγκομιδών κτλ. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να είμαστε ρεαλιστές στις αποφάσεις μας και να λάβουμε τις ε, αποφάσεις μας με τρόπο ο οποίος είναι εμπεριστατωμένος γιατί οι επιστημονικές ε, εμπειρογνωμοσύνες μπορούν να αλλάξουν από τη μια μέρα στην άλλη. Ο κύριος Ζουάου Φερέιρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω να κάνω δύο ή τρεις σύντομες παρατηρήσεις. Πρώτα απ' όλα, πιστεύω ότι το ψήφισμά μας δεν αντιμετωπίζει ορισμένα θεμελιώδη ζητήματα το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής, όπως αναφέρθηκε πολλές φορές, συνδέεται άμεσα με τη μεγάλη εξάρτηση που έχει ο κόσμος μας από τα ορυκτά καύσιμα και το υψηλό, υψηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα της οικονομικής μας και βιομηχανικής δραστηριότητας. Αυτό απαιτεί μια εγκάρσια αντιμετώπιση, μια οριζόντια αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων. Και σήμερα έχουμε ακόμα τεράστιες αντιφάσεις σε ό,τι αφορά τον πολιτικό λόγο και τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τη μια μεριά θέλουμε να παίξουμε ένα ρόλο ηγέτη για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, αλλά άλλες φορές, παράλληλα, πέραν των ασυναρτησιών της αγροτικής μας πολιτικής, εξακολουθούμε να είμαστε ενθου, ενθουσιώδεις υπέρμαχοι της κατάλυσης των φραγμών σε παγκόσμιο εμπόριο. Θέλουμε κοινέ πολιτικέ, όπω η κοινή αγροτική πολιτική. Θέλουμε όμω και συμφωνίε ελεύθερου εμπορίου που έχουν τεράστια επίπτωση στην κλιματική αλλαγή και πρέπει να αντιμετωπιστούν. Έχουμε την μετακίνηση των διαδικασιών παραγωγής, έχουμε τροποποίηση του τρόπου κατανάλωσης, έχουμε νέες μορφές παραγωγή που οδηγούν ουσιαστικά σε σημαντική αύξηση των ε, αερίων θερμοκηπίου. Υπάρχουν τεράστιες μεταφορές λοιπόν ενέργειας και πρώτων υλών σε παγκόσμιο επίπεδο και αυτό φυσικά συμβάλλει σημαντικά στην κλιματική αλλαγή. Η ανθρωπότητα αυτή αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή ένα πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Αλλά δεν είναι δυνατόν μέσα στο τρέχον οικονομικό σύστημα να βρούμε λύσεις για αυτό το πρόβλημα. Και πιστεύω ότι θα πρέπει λοιπόν να δούμε με πιο προσεκτικό τρόπο την αντιμετώπιση του θέματος αυτού. Δεν μπορούμε να βασιζόμαστε μόνο στους μηχανισμούς της αγοράς για να μπορέσουμε να βρούμε λύσεις στο πρόβλημα αυτό. Πιστεύω ότι η αποτελεσματικότητα των μηχανισμών της αγοράς για να μπορέσει να αντιμετωπίσει το σημαντικό αυτό πρόβλημα των εκπομπών είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να παραμείνει <clears throat> υπό εποπτεία. Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι αμφιβάλλουν και αιτιολογημένα για τη δυνατότητα του συνθήματος, συστήματος αυτού να αντιμετωπίσει την κλιματική αλλαγή. Αλλά εξάλλου η εφαρμογή αυτών των εργαλείων της αγοράς έχει και προβλήματα σε επίπεδο περιβάλλοντος και σε επίπεδο απασχόλησης. Μπορούν να προκύψουν διαφοροποιημένε συνέπειε για τι διάφορε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση και επομένω, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να λάβει υπόψη και αυτή την προβληματική ότι μπορούν να πληγούν με ορισμένε χώρε πολύ περισσότερο. Τέλο, όταν μιλάμε για μια διαφοροποιημένη υπευθυνότητα είναι χρήσιμο να λαμβάνουμε υπόψη ότι αυτή η έννοια θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί και μέσα στα πλαίσια της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδομένου ότι δεν έχουν όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης την ίδια ιστορική συμβολή στον τομέα των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακο. Υπάρχει μια τεράστια ποικιλομορφία μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να ληφθεί υπόψη στη συζήτηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο Σέργιο Μπελάτο έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κοιτάξτε, από το 99 είμαι εδώ στο Κοινοβούλιο και ειλικρινά σας λέω ότι ζηλεύω ορισμένους συναδέλφους ε, για τις βεβαιότητες που έχουν όσον αφορά ε, την διεξαγωγή ορισμένων μαχών. Ζηλεύω πολλούς συναδέλφους λοιπόν που στηρίζουν τις βεβαιότητές τους σε επιστημονικά στοιχεία που κατά την άποψή του είναι αδιαφυσβήτητα. Έχω διαβάσει πολλέ δημοσιεύσει από πολλού επιστήμονε και δεν έχω βρει ούτε και μία δημοσίευση που να μου δημιουργεί τη βεβαιότητα, την αδιαφυσβήτητη βεβαιότητα ότι η κλιματική αλλαγή σίγουρα συνδέεται, είναι ανθρωπογενού ε, προέλευση. Συνδέεται με τον άνθρωπο. Και το άλλα, να σα πω ότι πραγματικά ζηλεύω τη βεβαιότητα με την οποία ορισμένοι συνάδελφοι υποστηρίζουν, ε, υποστήριζαν τη θέση για την τρύπα του όζοντος. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή γνώμη είχε τρομοκρατηθεί τότε. Φοβόταν ο κόσμος να ε, ε, βγει στο δρόμο να κάνει μια βόλτα. Ότι θα ψηθεί δηλαδή από τον ήλιο λόγω της τρύπα του όζοντος. Εδώ και αρκετό καιρό δεν ακούμε τίποτα για το όζον και δεν ξέρω τι έγινε. Τι έγινε, πήγε κάποιο εκεί, ανέβηκε μια σκάλα και έβαλε ένα μπάλωμα και την έκλεισε τρυποτώζοντα. Αυτό έγινε. Υπάρχει, θέλω να πω, μία ε, καταστροφολογία. Και θα πρέπει να είμαστε αντίθετα πιο ρεαλιστές. Βεβαίω είναι σαφέ ότι πάντα υπεράσπιζα και ήμουν ένθερμος υποστηρικτής της ιδέας ε, της, διασφα... της για λόγου ανάγκη. Άρα λοιπόν Σίγουρα πρέπει να καταπολεμούμε τη ρήπανση, αλλά με αίσθημα ευθύνη. Άκουσα όμω ορισμένου συναδέλφου να κάνουν έτσι κάποιε ε, δηλώσεις ε, που πραγματικά ε, ήταν υπερβολικές χωρίς να καταλαβαίνουν καθόλου τι επιπτώσεις θα έχουν όλα αυτά σε ανθρώπινο επίπεδο, σε παραγωγικό επίπεδο, σε οικονομικό επίπεδο. Ορισμένες δηλαδή πρωτοβουλίες θεωρητικές αλλά που αν εφαρμοστούν θα έχουν καταστρεπτικά αποτελέσματα στις οικονομίες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανοίγοντας διάπλατα τις πόρτες σε ε, εισβολές άλλων χωρών που ήδη ασκούν αθέμητο ανταγωνισμό και ντάμπινγκ στην οικονομία της Ευρώπης. Επίσης, ε, πιστεύω ότι ακούω ότι θα πρέπει να χρηματοδοτήσουμε τις χώρες αυτές που ήδη ασκούν αθέμητο ανταγωνισμό. Αναφέρομαι στην Κίνα, στην Ινδία, στη Βραζιλία και χωρί καν να ξέρουμε αν αυτή αυτά τα κονδύλια θα χρησιμοποιηθούν για τη σωστή κατεύθυνση ή δεν θα χρηματοδοτήσουν ακόμα περισσότερο αυτό τον αθέμητο ανταγωνισμό που πλήττει την οικονομία μα. Λοιπόν, εάν εμεί συνεχίσουμε στηριζόμενοι σε αυτέ τι θεωρητικέ υποθέσει, συνεχίσουμε να επιβάλλουμε στην παραγωγική μας και στην οικονομική μας δραστηριότητα αυτούς αβάσταχτους, ε, αβάσταχτα εμπόδια, θα γίνει αυτό που έγινε και στη Γεωργία. Όπου αυτός που προστατεύει το περιβάλλον εξ ανάγκης, διότι ξέρει ότι εκεί ζει και εκεί δουλεύει. Από εκεί προσδοκά ένα καλύτερο μέλλον. Άρα, όπως σας είπα, εξ προστατεύει το περιβάλλον. Σε τελευταία ανάλυση θα οδηγηθούμε σε απερίμωση της υπαίθρου που θα οδηγηθεί σε εκφυλισμό και σε επιδείνωση της κατάστασης. Θα σταματήσω εδώ λοιπόν και σας λέω ότι δέχομαι πολύ ευχαρίστω την ε, πρόσκληση που είπε η κυρία Γκροστέτη, η οποία μας είπε το εξή, την έκκλησή της μάλλον. Ας βάζουμε εφικτούς στόχους και δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις έτσι ώστε η κοινή προσπάθεια να μας οδηγήσει σε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Γιατί αυτά τα οποία άκουσα σήμερα επανειλημμένα και το έχω ακούσει επανειλημμένα είναι δηλώσεις επί της αρχής, στηριζόμενες σε θεωρίες που δεν έχουν αποδειχθεί και που αύριο θα μας οδηγήσει σε αυτό ακριβώς που συνέβη και στην περίπτωση της τρύπας του όζοντος. Ότι θα καταλάβουμε δηλαδή ότι κάποιος μας περιπέζει και μας οδηγεί στο να ακολουθήσουμε λύσεις που συμφέρουν ορισμένους. Ας φροντίσουμε λοιπόν να είμαστε προσεκτικοί έτσι ώστε να δούμε τι γίνεται με, τις, ε, ε, ε, με την ενέργεια, αλλά ακούω ορισμένου περιβαλλοντολόγου έτσι και ακραίου που εκφράζει τη λύπη του για το γεγονό ότι χρησιμοποιούμε πάρα πολύ τα ορυκτά καύσιμα. Μην ξεχνάμε όμως τι γίνεται με τα πυρηνικά. Ε, όλα αυτά είναι, αν μη τι άλλο, αξιόπιστα. Τον ίδιο άνθρωποι έλεγαν τα, να χρησιμοποιούμε το ορεικτά καύσιμα και να μην καταφεύγουμε στην πυρηνική ενέργεια. Σας ευχαριστούμε. Βεβαίως ε, μίκρινε η τρύπα του όζοντος επειδή πλέον έχουν μειωθεί η χρήση των επικίνδυνων ουσιών που την προκαλούσαν. Για παράδειγμα, ό,τι περιείχε χρολοφρολάνθρακες. Και τώρα η Άζα Βέστλαντ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Κοιτάξτε, κατά την προεκλογική εκστρατεία, αναφέρομαι σε εκλογές του Ευρωκοινοβουλίου, συχνά ε, οι ψηφοφόροι μου έφεραν το ερώτημα και κυρίως ε, μέσω του blog μου στο διαδίκτυο μου έφεραν ερωτήματα που έχουν να κάνουν με το πάνελ για την κλιματική αλλαγή και με το γεγονό ότι ε, ε, οι, οι, απόψεις των, οι απόψεις τους και επικρίσεις τους δεν ακούγονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κοιτάξτε, θα έλεγα ότι σε γενικέ γραμμέ υπάρχει συμφωνία ανάμεσα στου πολιτικού και στου ερευνητέ ε, σε ολόκληρο τον κόσμο. Και στην προηγούμενη θητεία είχαμε καλέσει τους προσώπους του πάνελ των Ηνωμένων Εθνών που είναι υπεύθυνοι για το κλίμα και είχαμε θέσει μια σειρά από ερωτήματα. πήραμε ε, απαντήσεις ιδιαίτερα αξιόπιστες ε, και καλά επεξεργασμένες. Και εγώ λέω το εξής. Αυτά τα σωστά ερωτήματα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε και θα βρούμε τις σωστές απαντήσεις. Υπάρχει τώρα το εξής. Οι αλλαγές δεν, το, δεν επιβεβαιώνεται μόνο από την επιστήμη, αλλά και από την κοινή λογική. Ο καθένα μπορεί να δει την κλιματική αλλαγή. Η κλιματική αλλαγή ε, θα οδηγήσει σε ξηρασία, σε πλημμύρε σε ορισμένε περιοχέ του κόσμου, σε υπερθέρμανση και φαινόμενα τα οποία τα βλέπουμε καθημερινά. Νομίζω λοιπόν ότι Δεν μπορούμε να συνδέσουμε αυτά που μας λένε οι επιστήμονες με αυτά που, ε, που, γίνονται στην πράξη, με αυτά που βλέπουμε όλοι μας. Ε, εάν λοιπόν ε, οι φιλοδοξίες μας σε περιορίζονται στο 25% παρόλο που ήδη γνωρίζουμε ότι του στόχου του πετύχουμε μόνο αν φτάσουμε στο 50%, ε, τότε τι να πω, δεν ξέρω. Νομίζω ότι είναι σκανδαλώδης αυτή η συμπεριφορά τουλάχιστον να, να, να εβάλουμε στόχο το 40%. Σίγουρα πρέπει να αντιμετωπίσουμε ε, τους στόχους μας και να μην αφήνουμε ε, να μας παρασύρουν ε, αυτοί που δεν θέλουν ε, να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση κατάματα. Λοιπόν, προφανώς είμαι υπέρ πιο φιλόδοξων στόχων, αλλά συμφωνώ ταυτόχρονα και συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό με ε, το έγγραφο του Κοινοβουλίου. Αν στην Κοπεχάγη θέλουμε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία, τότε θα πρέπει να προσαρμόσουμε του στόχου μα με, με τα τελευταία επιστημονικά δεδομένα και τι τελευταίε επιστημονικέ μελέτε, τι πιο πρόσφατε. Λοιπόν, αυτά θα ήθελα να πω. Ε, οι εμπειρογνώμονε θα πρέπει να συνδεθούν στις διαπραγματεύσεις, να συμμετάσχουν. Αυτό θα ήταν κάτι το επιθυμητό. Το ψήφισμα ταυτόχρονα θα μπορούσε να αναφέρει πιο συγκεκριμένα τα ωφέλη ε, που θα μπορούσαν να προκύψουν για όλους. Αυτή λοιπόν η πτυχή θα μπορούσε να ξεκαθαριστεί καλύτερα. γνωρίζουμε ότι υπάρχει ευρεία συνένεση ανάμεσα στους επιστήμονες σε ολόκληρο τον κόσμο στο γεγονός ότι αυτό το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα σοβαρό. Γνωρίζουμε ταυτόχρονα ότι θα υπάρξουν σημαντικά οικονομικά ωφέλη εάν δράσουμε έγκαιρα. Εάν εμείς ως ε, ε, η Ευρώπη ε, είμαστε πορτοπόροι, θα είναι προς όφελος της ε, οικονομίας μας. Θα ήταν πραγματικά βλακώδες αν μετά, μέσα από όλα αυτά, μετά από όλα αυτά δεν μπορούμε να καταλάβουμε το μήνυμα το οποίο είναι σαφές. Βεβαίως υπάρχουν αντικρουόμενα συμφέροντα και το αντιλαμβανόμαστε. Αλλά δεν μπορούμε μόνο ε, να ε, ακούμε τους μεν και όχι τους δε. Θέλουμε να ωφεληθεί η κοινωνία σύνολό της. Άρα λοιπόν πρέπει να ακούσουμε όλα τα επιστημονικά στοιχεία. Ε, Ο Φίλιπ Ζουβάν έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Σαν νέος βουλευτής είμαι λιγάκι τρομοκρατημένος από ορισμένε παρεμβάσεις που έχω ακούσει. ανακαλύπτω μια συνέλευση η οποία αμφιταλαντεύεται ανάμεσα σε μια μεγάλη δυσπιστία γιατί δεν βασίζεται, δεν μπορεί να βασίζεται απόλυτα σε επιστημονικές γνώμες και από την άλλη μεριά μια πτέρυγα η οποία είναι απόλυτα πεπισμένη για την αξία αυτών των επιστημονικών θέσεων. Χρειαζόμαστε κοινή λογική και χρειαζόμαστε και κριτικό πνεύμα όμως. Παραδείγματο υπάρχουν συνάδελφοι που λένε ότι πρέπει να δούμε τι μας λέει η κοινή λογική. Η κοινή λογική πολλές φορές μας δίνει λαθασμένα αποτελέσματα. Νομίζουμε ότι γίνεται επίπεδη γιατί άμα την κοιτάξουμε μας φαίνεται επίπεδη. Σας δίνω τώρα ένα άλλο παράδειγμα της έλλειψης ρεαλισμού μέσα στη συζήτηση αυτή. Ορισμένοι συνάδελφοι είπαν ότι αν μειώσουμε το χρόνο εργασία, θα μειώσουμε και την αύξηση τη θερμοκρασίας. Ε, εντάξει, όλα μπορούμε να τα πούμε. Αν δίναμε και λιγότερα αντιβιωτικά, όχι μόνο δεν θα υπάρχει ρήπανση της χημικής βιομηχανίας, αλλά μειώνοντας και το προσδόκιμο επιβίωσης θα μειώναμε την ανθρωπογενή ρήπανση στον πλανήτη μας. Λοιπόν, μια τέτοια μορφή συζήτηση μα οδηγεί σε τελείω αντιρεαλιστικά συμπεράσματα. Να έρθω τώρα πιο συγκεκριμένα στο ψήφισμα. Το ψήφισμα αυτό το οποίο διάβασα όπως όλοι μας με μεγάλη προσοχή. Απαιτεί τις εξής τέσσερις παρατήρησεις. Μια γενική παρατήρηση είναι ότι δεν μπορούμε με την ευκαιρία μονάχα ενός ψηφίσματος δεν μπορούμε να αποφασίσουμε να ανατρέψουμε <clears throat> και να καταργήσουμε προηγούμενες δεσμεύσεις μας. Στο πακέτο ενεργείας κλίματος του είχε αποφασιστεί ο στόχος του 20% για τη μείωση των εκπομπών. Μετά από μια πολιτική συζήτηση. Ενώ εδώ πέρα βλέπω να εμφανίζεται ένα στόχος 40% που βγαίνει από κάποιο καπέλο. Γιατί 40%. Γιατί όχι 50, γιατί όχι 60. Είμαι ανοιχτός σε οποιαδήποτε συζήτηση. Απλώς θα ήθελα να ξέρω ότι αυτό το ποσοστό θα πρέπει να προέρχεται από μια επιστημονική έρευνα, κάτι που είναι πολύ πολύπλοκο, αλλά επίση και να προέρχεται από δημοκρατική συζήτηση, η οποία δημοκρατική συζήτηση έδωσε 20% Γιατί λέμε σήμερα 40%. Πιστεύω λοιπόν ότι γενικά το ψήφισμα δεν πρέπει να είναι ένα στοιχείο που να ανατρέπει δημοκρατικά ηλυμένες αποφάσεις. Τέσσερα στοιχεία τα οποία θα οδηγήσουν σε τέσσερις τροπολογίες. Καταρχήν, στο σημείο 2, <clears throat> όταν μας λέγεται ότι θα πρέπει να ζητήσουμε στις ε, βιομηχανικές χώρες να δώσουν το παράδειγμα και επίσης οι αναπτυσσόμενες χώρες να λάβουν υπόψη την ανάγκη να παρακολουθήσουν αυτή την αλλαγή. Οι τρει χώρε που αναφέρονται, η Κίνα, η Ινδία και η Βραζιλία, είναι οι χώρε που έχουν τη μεγαλύτερη αντίθεση στι δικέ μα θέσει και θέλουν να καταστρέψουν την ευρωπαϊκή οικονομία. Θέλω λοιπόν να υπάρξει μια διαφοροποίηση μεταξύ των αναπτυσσομένων χωρών που χρειάζονται βοήθεια, των αναδειωμένων χωρών και των χωρών που είναι άμεση ανταγωνιστές ευρωπαϊκής βιομηχανίας και που είναι κυρίως η Κίνα και η Ινδία. Λοιπόν, οι χώρες αυτές έχουν στόχοι που είναι διαφορετικοί από εμά. <clears throat> Επίσης, στο σημείο 3 μιλάμε για την ψαλίδα αυτή που πάει από 25-40%. Σας είπα ποια είναι η απόψή μου. Εγώ νομίζω ότι ο στόχος πρέπει να είναι 20% και όχι 40%. Η τρίτη μου παρατήρηση αφορά όλα αυτά τα θέματα που έχουν αντιμετωπιστεί από ορισμένου από εσά, αλλά που δεν έχει παρουσιαστεί στο ψήφισμα, επαρκώ είναι το θέμα τη προστασία τη βιομηχανία μα, δηλαδή του φόρου που πρέπει να εφαρμόσετε στα σύνορα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να έχουμε στόχου λοιπόν Στόχου για το περιβάλλον, αυτό είναι θετικό, αλλά δεν θα πρέπει αυτό να οδηγήσει σε αθέμητο ανταγωνισμό από την πλευρά βιομηχανιών που βρίσκονται σε τρίτες χώρε και που δεν έχουν τι ίδιε επιταγές προστασίας του περιβάλλοντος. Πρέπει να λάβουμε λοιπόν στα σύνορά μα κάποια μέτρα, τα οποία εναπόκειται και για μένα στους εμπειρογνώμονε, για να αντιμετωπίσουμε την δυνητικά αθέμητη μορφή ανταγωνισμού. Τέλο έρχομαι στο σημείο 8. Στο σημείο 8 λέει ότι η συλλογική συνεισφορά τη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 30 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίω μέχρι το 2020. Τώρα εγώ δεν ξέρω αν πρέπει να είναι 30, 40, 50. Δεν με ενδιαφέρει ποιο είναι το ποσό, τι θα πρέπει να προκύψει. Εγώ νομίζω 20 δισεκατομμύρια που να χρησιμοποιηθούν σωστά, παρά 30 δισεκατομμύρια τα οποία μπορεί να κατασπαταλεθούν. Ευχαριστώ λοιπόν κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ αγαπητέ συνάδελφε. Νομίζω όμως ότι αυτό που αναφέρατε δεν είναι απόλυτα επακριβές. Αν δείτε την αιτιολογική σκέψη ΔΕΛΤΑ παραδείγματο χάρη, παραμένουμε στις αποφάσεις οι οποίες ελήφθησαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση 20% μέχρι το 2020 και στην περίπτωση που θα μπορούσε να προκύψει μια συμφωνία στην Κοπεχάγη τονίζαμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να προχωρήσει περισσότερο μέχρι το 30%. Χωρίς ο μικρόφωνο μιλητής. Εσείς αναφέρεστε στο άρθρο 3, το οποίο απλώς αναφέρει αυτό το οποίο είπε το πάνελ για την κλιματική αλλαγή, η Επιτροπή για την κλιματική αλλαγή, συγγνώμη, για το 25 μέχρι 40% που είναι αυτό το οποίο είναι απαραίτητο σύμφωνα με τους επιστήμονες να γίνει μέσα στις βιομηχανικές χώρες για να επιτευχθεί ο στόχος. Απλώς θέλω να σας ε, αναφέρω ότι στο κείμενο δεν υπάρχει κάποια... Είπατε ότι δεν υπάρχει κάποιο στο κείμενο αυτό το θέμα του 40%. Η Λίντα Μακέβεν τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς, θα ήθελα να απαντήσω στον Ιταλό συνάδελφο από το ΕΛΚ που μίλησε για το Όζον ότι θα μπορούσε η Γραμματεία να του στείλει τη Διεθνή Συμφωνία για την αντιμετώπιση της τρύπης του Όζοντος για να δει ότι καταφέραμε να επιλύσουμε τα προβλήματα και αυτό θέλουμε να κάνουμε και τώρα. Θέλουμε να έχουμε μια Διεθνή Συμφωνία που θα αντιμετωπίσει ένα πραγματικό πρόβλημα που έχουν αντιμετωπίσει οι επιστήμονες. Και στο συνάδελφο που μόλις μίλησε, δεν μπορούμε τώρα να αναθεωρήσουμε τα επιστημονικά στοιχεία και να αναθεωρήσουμε και τις αποφάσεις που έχουμε ήδη λάβει. Στην Κοπενχάγη το βασικό θα είναι να μπορέσουμε να βάλουμε και άλλες χώρες στον χώρο και το κλειδί εδώ θα είναι η εκβιομηχανισμένες χώρες να πάνε στην Κοπενχάγη με μια αξιόπιστη πρόταση. Και πρώτον να έχουμε ένα πακέτο μέτρων για μετρίαση των συνεπειών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις εκβιομηχανισμένες χώρες, κάτι που το κάναμε πέρυσι με το πακέτο που αναφέρει μείωση τουλάχιστον 20% και μείωση 30% αν υπάρξει διεθνή συμφωνία και συνένεση. Τώρα, το 40% θα είναι δύσκολος στόχος. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή στο Συμβούλιο ότι υπάρχουν ε, και φωνές που ζητούν να αλλάξει ο στόχος του 20%. Οπότε, πρέπει να έχουμε υψηλούς στόχους στην Κομεχάγη. Γι' αυτό βάζουμε 25-40% αν και θα θέλαμε και το 40%. Πάντως αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να ξανανοίξουμε θέματα που έχουν ήδη συμφωνηθεί, ήδη συμφωνήθηκαν πέρυσι, όπως η εμπορία εκπομπών κτλ τώρα. Το σημαντικό είναι η Κοπενχάγη και είναι σημαντικό τα θέματα χρηματοδότησης να αποφασιστούν γιατί αυτά είναι που θα καθορίσουν την έκβαση της Κοπενχάγης και εκεί όλα τα μάτια θα είναι στραμμένα προς την Κοπενχάγη. Ο κύριος Παρόσο μας είπε ποιο είναι το πακέτο την προηγούμενη εβδομάδα. Γνωρίζουμε ότι οι οικονομικές συνθήκες είναι δύσκολες και όλες οι χώρες αντιμετωπίζουν προβλήματα σήμερα. Όμως χρειαζόμαστε ένα αξιόπιστο πακέτο για να μπορέσουμε να εμπλέξουμε και άλλες χώρες. Γιατί αν δεν εμπλέξουμε και άλλες χώρες δεν θα καταφέρουμε να μειώσουμε τις εκπομπές άνθρακα. Γιατί αν μέχρι το 2050 όλες οι υπόλοιπες χώρες μειώσουν τις εκπομπές στο μηδέν, αλλά όχι η Ινδία και η Κίνα, τότε πάλι δεν θα μπορέσουμε να επιτύχουμε τους στόχους μας. Άρα πρέπει να έχουμε σαφείς προτάσεις. Πρέπει να είμαστε αξιόπιστοι. Πρέπει να αναλάβουμε και τις δικές μας ευθύνες. Πρέπει να βρούμε χρηματοδότηση πέρα από αυτή που ήδη έχουμε υποσχεθεί. Δεν μπορούμε να πάμε στις αναπτυσσόμενες χώρες και να τους πούμε ότι θα σας δώσουμε χρήματα από αυτά που σας είχαμε ήδη υποσχεθεί στο Glen Eagles πριν από τρεις, τρία χρόνια, τότε δεν θα είμαστε αξιόπιστοι. Πρέπει να βρούμε επιπλέον χρηματοδότηση πέρα από την κλασική αναπτυξιακή βοήθεια. Και πρέπει να βρούμε τρόπους αξιόπιστης και μετρήσιμης αλλαγής στα θέματα της αντιμετώπισης κλιματικής αλλαγής. Έχουμε τους στόχους της χιλιετίας, αλλά ήδη γνωρίζουμε ότι αρκετά κράτη-μέλη δεν έχουν συμμορφωθεί με τους στόχους τους. Και Παρακαλώ συνάδελφοι, επικεντρωθείτε στο ψήφισμα και στην Κοπενχάγη. Αν θέλουμε να ακουστεί η φωνή του Κοινοβουλίου, πρέπει να επικεντρωθούμε σε 4-5 σημεία βασικά. Δεν μπορούμε να μιλάμε περί ανέμων και υδάτων. Πρέπει να δείξουμε ακριβώς ποια είναι τα στοιχεία που πρέπει να αποτελέσουν κομμάτι της συμφωνίας. Από εκεί και πέρα υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούν να ακολουθήσουν αποψήλωση, offsetting κτλ. Όμως τώρα ας επικεντρωθούμε στα βασικά. Και κάποιοι από εμά θα πάμε στην Ουάσιγκτον. Ας συζητήσουμε με τους εταίρους μας ε, της ΣΥΠΑ. Και έχουμε δει και κάποια ενθαρρυντικά μηνύματα όπως για παράδειγμα σήμερα που διαβάζουμε στους New York Times ότι κάποιες σημαντικές πολυεθνικές εταιρείες συμφωνούν με τη λήψη μέτρων και μάλιστα έφυγαν και από το εμπορικό επιμελητήριο των Ηνωμένων Πολιτειών επειδή αυτό αντιτίθεται στα μέτρα. στα μέτρα όσον αφορά την εμπορία των εκπομπών. Άρα, διαπιστώνουμε ότι το να υπάρχει αξιόπιστη σαφής νομοθεσία είναι σημαντική για την οικονομία και όσο περισσότερο καθυστερούμε τόσο πιο δύσκολο θα είναι τα πράγματα. Τέλος, επαναλαμβάνω, ας επικεντρωθούμε στα βασικά. Ευχαριστώ. And finally, Mario Πρόεδρε, δεν ήθελα να πάρω το λόγο. Ε, αλλά να σας πω την αλήθεια, επειδή ε, ε, εγώ παρακολουθώ ιδιαίτερα προσεκτικά τη συζήτηση για την Κοπενχάγη. Αντιλαμβάνομαι. Για στιγμή έχουμε πρόβλημα διαμηνίας, λέει ο πρόεδρος. Μ' ακούτε τώρα. Υπάρχει ένα πρόβλημα με την διερμηνία. Ναι, ωραία. Εντάξει, δεν σε ακούω. Λοιπόν, έλεγα, Πρόεδρε, ότι δεν ήθελα να πάρω το λόγο, αλλά μετά ορίμασε η ιδέα. Να κάνω μια πολύ σύντομη παρέμβαση σε σχέση με τη συζήτηση που όπως διαμορφώθηκε σήμερα. Συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό με αυτά τα θέματα ε, της Κοπενχάγης και με τα αποτελέσματα. Και περιμένω πολλά από τα αποτελέσματα. Κοιτάξτε, στην Κοπενχάγη πρέπει να πάει αυτό το έγγραφο το οποίο αποτέλεσε αντικείμενο συζήτηση σήμερα το πρωί και που νομίζω ότι περιέχει πάρα πολλά θετικά σημεία. Και ίσως δεν το διαβάσαμε αρκετά καλά. Ίσως η ορολογία μας ξεφεύγει, δηλαδή αφορά οι δήμονες και όχι οι ανθρώπους που δεν είναι εξοικειωμένοι με αυτούς τους όρους και που για πρώτη φορά εδώ στο Κοινοβούλιο ασχολούνται με ένα τέτοιο πρόβλημα. Όπως το κλιματική αλλαγή που βεβαίως επηρεάζει όλους και μας αφορά όλους. Να σας πω ότι με τη μακροχρόνια μου εμπειρία ε, ως υπεύθυνο για τη γεωργία στη, χώρα μου, στη, στην περιοχή μου και βλέποντας το θέμα της αποψήλωσης, βλέπω πραγματικά ε, αποτελέσματα, βλέπω τι γίνεται, βλέπω ε, την αποψήλωση, βλέπω την περίμωση μάλλον. Ε, ένα πρόβλημα το οποίο θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Ε, και την αποψήλωση των δασών. Εμεί εργαστήκαμε πολύ προ την κατεύθυνση ανανεώσιμη ενέργεια και ήδη τα προγράμματα ε, τη ανάπτυξη πέθρου προβλέπουν για τις επιχειρήσεις μόνο παρεμβάσεις σε επίπεδο ανανεώσιμων ενεργειών. Αλλά βέβαια, εδώ που πρέπει να κάνουμε προσπάθεια είναι το θέμα του του ανταγωνισμού. Και θα πρέπει και στην Κοπεχάγη να υπογραμμιστεί το γεγονός αυτό. Ότι ορισμένε δηλαδή αναδυόμενε οικονομίες, και το είπαμε πολλοί συνάδελφοι, να μην επαναλάβω εδώ τα ίδια, η Κίνα, η Ινδία και άλλοι. Με τη στάση τους πρέπει να δούμε τι γίνεται. Ε, Λαμβάνοντα υπόψη και με την κατάσταση ορισμένων επιχειρήσεων. αυτά συμβαίνουν στην πράξη, δεν είναι θα συμβούν. Το λέω, ε, πρόεδρε, δεν είναι αβάσιμη φόβη αυτή. Έχουν γίνει μελέτες, υπάρχουν στοιχεία. Αυτά τα πράγματα ήδη συμβαίνουν. Ακριβώς γιατί ε, στις, φεύγουν από περιοχές όπου αποφάσισαν να μην δράσουν, για να αντιδράσουν σε αυτήν την κατάσταση. Όλα αυτά βεβαίω και προκαλούν ανησυχίε. Ανησυχίε που είχα κι εγώ. Και που μεγάλωσαν ακόμη περισσότερο σήμερα, ακούγοντα ε, του συναδέλφου και τι παρεμβάσει του. Θα σταματήσω εδώ. Σας ευχαριστώ και επαναλαμβάνω. Αυτό που με ανησυχεί είναι το θέμα του ανταγωνισμού. Ευχαριστώ πολύ. Έχει κλείσει λοιπόν η συζήτηση αυτή, η οποία ήταν πλήρης και ενδιαφέρουσα. Νομίζω ότι παρουσιάστηκε όλο το φάσμα απόψεων της Επιτροπής μας. Υπάρχει λοιπόν αυτή η διάσκεψη η οποία θα λάβει η χώρα. Ο στόχος της είναι η μείωση των εκπομπών αεροθερμοκηπίου και αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει η συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό αντανακλάται και στο ψήφισμα, σε αυτή την προσπάθεια και η αίτηση προς τις άλλες πλευρές να πράξουν τα αντίστοιχα. Δεν υπάρχει περίπτωση η Ευρώπη από μόνη της να σταθεροποιήσει το παγκόσμιο κλίμα. Χρειάζεται παγκόσμια συνεργασία. Προθεσμία για τις τροπολογίες 1η Οκτωβρίου 6 ώρα το απόγευμα, αύριο το βράδυ δηλαδή. Μέχρι αύριο το απόγευμα λοιπόν στις 6 ώρα θα πρέπει να κατατεθούν οι τροπολογίες σε σχέση με το ψήφισμα για να μπορέσουν να προλάβουν να μεταφραστούν κιόλα. Αγαπητοί συνάδελφοι λοιπόν μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο σημείο το οποίο συνάπτεται βέβαια με το προηγούμενο. Θέλουμε να καταθέσουμε μια προφορική ερώτηση προς την Κομισιόν και προς το Συμβούλιο Και με τον τρόπο αυτό μπορούμε να προετοιμάσουμε τη συζήτηση στην Ολομέλεια που θα κλείσει με το ψήφισμα το οποίο έχουμε καταθέσει. Έχετε το κείμενο της προφορικής ερώτησης σε όλες τις γλώσσες και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν έχετε κάποιες παρατηρήσεις ή σχόλια για το κείμενο αυτό. Κυρία Γκροστέτ. Ναι, είναι απόλυτα ε, σύμφωνο με αυτά τα οποία ελέγξαν σε σχέση με το ψήφισμα. Να πω το εξή. Ε, στην, στην πρώτη τελευταία παράγραφο που προτείνεται αυτή η ψαλίδα από 25-40%. Από πού προκύπτει. Εγώ είπα ότι ψηφίσαμε το πακέτο ενέργεια και κλίμα και όσοι ήμασταν στο προηγούμενο κοινοβούλιο θα θυμηθούμε το πόσο δύσκολα τα πράγματα και το πόσο είχαμε ανησυχήσει όλοι γιατί φοβόμασταν δεν θα καταλήξουμε πουθενά. Ε, γιατί στο πακέτο ε, ορίζαμε τις φιλοδοξίες μας και τις δεσμεύσεις μας για τη διάσκεψη Κοπεχάγης. Μείον 20% μέχρι το 2020 και μείον 30% αν έχουμε συμφωνία διεθνή, ικανοποιητική. Τώρα αρχίζουμε να μιλάμε για 20-40%. Τι να πω. Πολλοί είναι αυτοί στην ομάδα μου που δεν πρόκειται να το δεχτούν. Δηλαδή ζητάμε να σεβαστούμε τις δεσμεύσεις του πακέτου ενέργεια για κλίμα που ψηφίσαμε πριν από 9 μήνες. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι στο πακέτο του κλίματος υπάρχει και ο μακροπρόθεσμος στόχος. Δηλαδή, είμαστε δεσμευμένοι για το 20% στην περίπτωση συμφωνίας στην Κοπεχάγη και για το 30% αυτά είναι τα δεδομένα στοιχεία αλλά νομίζω ότι στη συζήτηση αυτή και στο, στην απόφαση του Συμβουλίου αναφέρθηκε και η δυνατότητα να προχωρήσουμε σε πιο φιλόδοξους στόχους ακόμα και 80% μέχρι το 2050 από την πλευρά της βιομηχανίας. Το ερώτημα είναι γιατί δεν θα πρέπει το Κοινοβούλιο να θέσει αυτό το ερώτημα στην Κομισιόν και στο Συμβούλιο. Κύριος Λίζε, θέλω να κάνω μια πρόταση που θα μπορούσε ίσως να επιλύσει το πρόβλημα αυτό. Νομίζω ότι η ψαλίδα αυτή το 25 με 40% είναι κάτι που προέρχεται από το Κοινοβούλιο και από τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την χάνει την υποστήριξή τους, είναι τα αποτελέσματα της διάσκεψης του μπαλή. Αλλά δεν υπάρχει ακόμα παγκόσμια συνένεση για τα θέματα αυτά. Γι' αυτό πρέπει να το συζητήσουμε ακόμα στην Επιτροπή μας και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σαν σύνολο. Εγώ πιστεύω ότι αυτά που αναφέρονται στο άνω άκρο της ψαλίδας είναι προϊόντα της ε, συνδιάσκεψης του Μπαλί και των θέσεων του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Δεν μπορεί κανεί να θεωρήσει ότι υπάρχει βέβαια συνένεση για τα θέματα αυτά. Νομίζω θα πρέπει να επανέλθουμε στην, στο άνω όριο τη ψαλίδα σε ένα μεταγενέστερο χρονικό σημείο. Μακίβαν. Κοιτάξτε, δεν πρέπει να συγχαίουμε τα πράγματα. Είναι αλήθεια ότι πέρυσι συμφωνήσαμε 20, ε, στο 20-30% και ότι υπάρχει αυτό στο νομοθετικό πακέτο. Αλλά εδώ μιλάμε για κάτι διαφορετικό. Μιλάμε για αυτό το οποίο είπε η Διεθνή Επιτροπή ότι χρειαζόμαστε. Επαναλαμβάνουμε δηλαδή τα επιστημονικά δεδομένα, αυτά που είπαν οι επιστήμονε. Δηλαδή, κοιτάξτε, αν το πείτε πολιτικά από την άψη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, που λέμε ότι πραγματικά το 20% δεν είναι αρκετό, τώρα έχουμε και την επιβεβαίωση από του επιστήμονε. Ο 30% δηλαδή είναι το ελάχιστο. Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω με κάτι το οποίο στην ουσία ε, αγνοεί ε, τα γεγονότα τα οποία φαίνονται και μέσα από την τέταρτη έκθεση αξιολόγηση. Ε, παρακαλώ λοιπόν του συναδέλφου να μην αγνοούν τα γεγονότα. Ναι, βεβαίω, συμφωνήσαμε σε μία δέσμη που είπαμε 20-30%, αλλά εδώ είναι κάτι τελείω διαφορετικό. Ο Να διευκρινίσω ότι ο στόχος του 25% και του 40% αφορά όλες τις βιομηχανοποιημένες χώρες. Αυτό βρίσκεται μέσα στα συμπεράσματα του Μπαλί. Ήταν η έκθεση του IPCC, του πάνελ για την κλιματική αλλαγή και έχει ήδη εγκρίνει το κοινοβούλιο μας το στόχο αυτό που περιλαμβάνει και το 40% για τις βιομηχανοποιημένες χώρες. Από την άλλη μεριά υπάρχει την Ευρώπη ο στόχος του 20 με 30%. Το 25 με 40% είναι αυτά τα οποία πρότεινε το Διεθνές Πάνελ για την Κλιματική Αλλαγή, ενεκρίθησαν στον Πάλι, στη διάσκεψη του Μπαλί, ενεκρίθησαν και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επίση. Επομένω, επαναλαμβάνουμε κάτι που έχει ήδη εγκρίνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο παρελθόν. Θα πρέπει να είναι σαφέ σε όλου. Monsieur le Président, je voulais revenir simplement sur le document que j'ai fait distribuer. Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει το έγγραφο που σας διένυμα. Τα αποτελέσματα της διάσκεψης στην οποία είχα αναφερθεί προηγουμένως. Σύμφωνα με αυτό, 91% των συμπολιτών μας θεωρούν ότι ο στόχος πρέπει να είναι 25 με 40% ή ακόμη μεγαλύτερος. Και 62% από αυτούς πιστεύουν ότι ο στόχος πρέπει να είναι 25 με 40% και το υπόλοιπο πάνω από 40% μέχρι το 91%. Δεν πρέπει να είμαστε αφελείς, παρόλα αυτά όμως υπάρχει συγκεκριμένη επιστημονική συνένεση και εκεί πρέπει να βασιστούν και οι πολιτικές μας. Καταλαβαίνω ότι μερικοί συνάδελφοι μπορεί να μπερδεύουν τις, ε, τους δικούς τους πόθου πόθους με τα πραγματικά στοιχεία. Όταν ε, ε, αναπαραπέμπουν σε επιστημονικές απόψεις που εκφράζονται ομόφωνα, δεν ε, αναφέρονται στην πραγματικότητα. Αν πάρω για παράδειγμα την άποψη ορισμένων επιστημόνων, ορισμένων από αυτούς που αναφέρονται σε αυτά τα στοιχεία. Ναι, υπάρχουν αυτέ οι απόψει, αλλά υπάρχουν και άλλε απόψει επιστημόνων που μιλούν για το διαμέτρο αντίθετο. Εμεί λοιπόν στο Κοινοβούλιο φτάσαμε σε ένα σημείο ισορροπία. Το οποίο θα πρέπει να το διατηρήσουμε. Μιλήσαμε για 20% που ήδη προήλθε μετά από μακροσκελής διαπραγματεύσεις και πολιτική συμφωνία να ε, ενισχύσουμε το κείμενο παραπέμποντας το μέλλον ε, να ενισχύσουμε το κείμενο παραπέμποντας σε, περισσότερα, σε υψηλότερα ε, ποσοστά, τα οποία δεν έχουν προκύψει από καμία συμφωνία, νομίζω ότι δεν είναι καθόλου σωστή τακτική. Νομίζω λοιπόν θα πρέπει να παραμείνουμε σε αυτή τη συμφωνία ε, σε αυτό το ποσοστό στο οποίο κατέληξε το, στο Κοινοβούλιο μετά από μακροσκελής διαπραγματεύσεις και συμφωνίες. Εγώ δεν είμαι, δεν προσωπώ τη βιομηχανία, ούτε τα συμφέροντά τους. Απλά και μόνο ζητώ να σεβαστούμε την πολιτική συμφωνία στην οποία καταλήξαμε πριν από ένα χρόνο μόλις, εδώ στο Κοινοβούλιο. Ε, ε, Ευχαριστώ. Ένα πράγμα πρέπει να θυσιάσουμε την οικονομία μας για το 40%. Κοιτάξτε, όσον αφορά τα επιστημονικά δεδομένα, νομίζω ότι έχουμε ακούσει αποκλίνουσες απόψεις και συμφωνώ με τον κύριο Ζουβάν ότι ναι μεν η ανθρώπινη δραστηριότητα δεν είναι αμεληταία, όμως ζούμε και ένα ζωντανό πλανήτη ο οποίος δημιουργεί πόρους κτλ. κτλ. Ας το λάβουμε υπόψη μας αυτό. Γιατί Γρυλανδία ονομάζεται Γρυλανδία, Greenland στα αγγλικά, γιατί κάποτε ήταν πράσινη. Οπότε ας μην τα μετατρέπουμε όλα σε δράμα για την ανθρωπότητα. Άλλους δύο μιλητές έχω. Μπάλτσιο. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Νομίζω ότι θα πρέπει να καταλήξουμε σε μία απόφαση. Εδώ έχουμε την προφορική ερώτηση προ το Συμβούλιο. Πού θα στηριχθούμε, σε επιστημονικά στοιχεία ή σε σφιγμομετρήσεις. Η σε σφιγμομετρησει η αποψη μου είναι και από ό,τι γνωρίζω έτσι έχουν τα πράγματα. Εάν Ε, θα πρέπει να, ε, ε, πάντα στις, στις, στις ερωτήσεις μας την πρέπει να στηρίζουμε σε επιστημονικά στοιχεία. Λοιπόν, ρωτώ, 5, 10, 20, 30, 40, ποιο ποσοστό υποστηρίζουμε. Κοιτάξτε, κάποιο που δεν ξέρει, έτσι ο απλός πολίτης ακολουθεί τη, τη μέση τομή, γιατί ε, θεωρεί ότι δεν έχει τα κατάλληλα στοιχεία. Ε, άρα λοιπόν οι συμμετρήσει είναι ενδιαφέρουσε, αλλά δεν νομίζω ότι ε, εκεί πρέπει να στηριζόμαστε όταν παίρνει μια απόφαση. Ζέμπα. Εγώ θα ήθελα να εκφράσω την άποψη ότι εδώ δεν νομίζω ότι εμείς μιλάμε για πραγματικά γεγονότα. Μιλάμε για προεκβολές στο μέλλον. Μιλάμε για εκτιμήσεις. Όλα αυτά είναι προβλέψεις και η έκθεση του IPCC αναφέρεται του πάνελ για την κλιματική αλλαγή αναφέρεται σε μια πιθανότητα ότι αυτά τα πράγματα θα είναι πραγματικότητα με μια συγκεκριμένη πιθανότητα. Δεν μπορούμε να τα θεωρήσουμε ως επιστημονικά εδρεωμένα ότι αυτά τα πράγματα θα είναι έτσι ακριβώς στο μέλλον. Έχουμε απλώς μοντέλα τα οποία προβλέπουν κάτι με μια ορισμένη πιθανότητα. Εγώ πιστεύω όπως ο Λίζε ότι εμείς θα πρέπει να συνεχίσουμε να έχουμε το, την εντολή διαπραγματεύσεως που είχαμε από το παρελθόν, από το πακέτο για την κλιματική αλλαγή και να το δούμε το 40% στη συνέχεια. Ευχαριστώ. Εγώ πρέπει να ομολογήσω ότι ούτε και εγώ ήθελα να μιλήσω σε αυτή τη συζήτηση. Παρ' όλα αυτά μιλάω, αφού άκουσα τι απόψει που διατυπώθηκαν. Δεν ξέρω ποια είναι η θέση στι δικής σα χώρε. Στην Πολωνία όμω ήταν πολύ δύσκολο να μπορέσουμε να πείσουμε τον κόσμο να υποστηρίξει το στόχο του 20%. Η χώρα μας ακόμα προσπαθεί να σηκωθεί και να σταθεί στα πόδια της μετά από το παρελθόν και το σύστημα που ισχύει εκεί πέρα. Είναι πολύ δύσκολο για μια χώρα σαν και εμάς που δεν έχουμε αναπτυγμένη βιομηχανία να επιτύχουμε αυτούς τους στόχους. Μπορεί κανείς να γράψει 80%, 100%, οτιδήποτε θέλει, όπως προτείνουν ορισμένοι συνάδελφοι. Στην πράξη όμως πρέπει να δούμε τι είναι εφικτό. Θα πρέπει να παραμείνουμε προσγειωμένοι. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να περισσώσουμε τις ε, βιομηχανίες στην Ευρώπη γιατί αν έχουμε ποσοστά τα οποία βρίσκονται στο άνω άκρο της ψαλίδας, το αποτέλεσμα είναι ότι οι βιομηχανίες μας θα πάνε στην Αφρική, σε άλλα μέρη του κόσμου που δεν υπάρχουν τέτοιου είδους περιορισμοί στην εκπομπή αερίων θερμοκηπίου. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να εξασφαλίσουμε την ισορροπημένη μια ισορροπημένη απόφαση. Ναι, θα πρέπει να ζητήσουμε να έχουμε μια αηφόρο ανάπτυξη, αλλά όχι πράγματα τα οποία είναι ανέφικτα. Ίσως είναι απαραίτητο να κοιτάξουμε και πάλι το κείμενο. Προσεκτικά λέει ο πρόεδρος. Τι λέει το κείμενο. Αναφερόμαστε σε αυτά τα οποία είπε το Διεθνές Πάνελ για την κλιματική αλλαγή που είναι ένας φορέας του ΟΗΕ και στον οποίο συμμετέχουν όλες οι χώρες μας και ο φορέας αυτός λέει ότι θα πρέπει να υπάρξει μείωση 25 με 40% σε σχέση με το 1990 σε όλες τις βιομηχανικές χώρες, όχι στην Ευρώπη, συγκεκριμένα, αλλά σε όλες τις βιομηχανικές χώρες. Αυτό λέει η πρόταση αυτή. Είναι μια κατεύθυνση και θέτουμε επί τη βάση αυτής της κατεύθυνσης το ερώτημα προς τη Κομισιόν και το Συμβούλιο τι θα γίνει λοιπόν ώστε να παραμείνουμε στα πλαίσια των προτάσεων των εμπειρογνωμόνων. Αυτό δεν σημαίνει ότι η Πολωνία μόνη της ή κάποια άλλη χώρα μόνη της θα πρέπει να βρεθεί στο άνω άκρο αυτής της ψαλίδας. Λέμε ότι θα πρέπει να δούμε πώς το Συμβούλιο ή η Κομισιόν μπορούν να αντιδράσουν στις προτάσεις των εμπειρογνώμων. Τώρα μπορεί κανείς να συμφωνεί ή να διαφωνεί με τους εμπειρογνώμονες. Δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας οδηγήσει τώρα σε αντιπαραθέσεις. Νομίζω ότι έχουμε τους επιστήμονες οι οποίοι δίνουν κάποια ε, πορίσματα τα οποία πιστεύω ότι πρέπει γενικά να τα λαμβάνουμε υπόψη. Μπορεί κανείς να έχει και μια διαφορετική άποψη άμα θέλει. Αυτό είναι δικαίωμά του. Έχουμε τρεις ακόμα που θέλουν να λάβουν το λόγο. Ο Πέτερ Λίζε και θέλει να λάβει το λόγο στο τέλος. Κυρία Βάις Γκέρμπερ και κύριο, κύριος Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχετε πράγματι δίκιο. Η προφορική αυτή ερώτηση αναφέρεται σε μια ψαλίδα που αφορά την πρόταση του πάνελ για την κλιματική αλλαγή, τις τέσσερις έκθεσεις αξιολόγησης του πάνελ για την κλιματική αλλαγή. Καταλαβαίνω όμως και τα επιχειρήματα ε, ορισμένων χωρών. Και γι' αυτό ίσως είναι σωστή η πρόταση του κ. Ζέμπερ να διαγράψουμε το άνω άκρο της ψαλίδας. Η δική μου άποψη είναι ότι προτού φτάσουμε στο 40% θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι προϋποθέσεις με τις οποίες όχι μόνο τα άλλα κράτη-μέλη, αλλά και τα άλλα κράτη σε παγκόσμιο επίπεδο θα δεσμευτούν για μία μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακος. Τουλάχιστον λοιπόν θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι τα μεγάλα βιομηχανικά κράτη να το πράξουν αυτό. Επομένως δεν έχει νόημα εμείς να <clears throat> προσπαθήσουμε να μειώσουμε τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακος, γιατί από μόνοι μας δεν μπορούμε να αλλάξουμε και να τροχοπεδίσουμε την κλιματική αλλαγή χωρίς τη συμμετοχή των άλλων μεγάλων χωρών του κόσμου. Ήταν σωστή η τελευταία σας παρατήρηση ότι αυτό είναι μια αναφορά στην έκθεση του IPCC. Εγώ πάντως <clears throat> πιστεύω ότι θα πρέπει να έχουμε μια σταδιακή προσέγγιση. Αν λοιπόν τα άλλα κράτη είναι έτοιμα να προχωρήσουν και αυτά σε βήματα, ίσως δεν πρέπει να διαγράψουμε αυτό το στόχο, αλλά να το κρατήσουμε κάτω από ορισμένε προϋποθέσεις. Ευχαριστώ. Ε, θα σας ε, έκανα μια διάλεξη για το γιατί ονομάζεται η Γρυλανδία Γρυλανδία. Σίγουρα δεν ονομάζεται έτσι επειδή κάποτε ήταν πράσινη. Αν θέλετε μπορώ να σας ε, το διευκρινίσω περαιτέρω. Τώρα, η συζήτηση για το 25 και το 40% κατά τη γνώμη μου δεν είναι η κατάλληλη συζήτηση αυτή τη στιγμή συζητάμε για κάποιες ώρες, αλλά δεν έχουμε μπει ούτε στις ερωτήσεις ούτε στο ψήφισμα. Αυτή τη στιγμή δεν πρέπει να αναθεωρήσουμε πράγματα που έχουμε αποφασίσει. Αυτό που κάνουμε είναι να επαναλάβουμε πράγματα που έχει ξαναπεί και το Κοινοβούλιο στο παρελθόν. Και η διατύπωση που χρησιμοποιούμε είναι η ίδια που είχε χρησιμοποιηθεί και στο παρελθόν. Τίποτα δεν υπάρχει καινούριο εδώ. Είναι αυτά που είχαν αναφερθεί στο παλι και τα οποία έχουμε υιοθετήσει αρκετές φορές. Αυτές είναι και οι πληροφορίες που έχω και εγώ πάρει από τη Γραμματεία στις 11 Μαρτίου 2009 στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου χρησιμοποίησαμε ακριβώς αυτή τη διατύπωση η οποία αναφέρεται και στην προφορική ερώτηση. Αυτό λοιπόν ήταν ένα ψήσιμο το οποίο ενεκρίθη με μεγάλη πλειοψηφία στο, στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τώρα το ερώτημα είναι αν θέλουμε να επαναλάβουμε αυτή την ε, διατύπωση ή αν θέλουμε να έχουμε μία άλλη αντιμετώπιση. Δεν ξέρω τώρα αν θα ήταν ε, πρέπον δύο μήνες πριν από την Κοπεχάγη να αλλάξουμε πορεία πλεύσης. Σας παρακαλώ λοιπόν να διαβάσετε αυτή την πρόταση προσεκτική, αναφέρεται σε όλες τις βιομηχανικές χώρες στον κόσμο και παραπέμπει στο γεγονός ότι το πάνελ για την κλιματική αλλαγή του ΟΗΕ είχε διατυπώσει αυτό το αίτημα. Λοιπόν, δεν είναι απλώς μια αίτηση, δεν σημαίνει ότι εμείς δεχόμαστε να, να διαγράψουμε την ε, απόφαση του πακέτου για την, κλιμα, κλιματική αλλαγή και την ενέργεια. Νομίζω λοιπόν ότι είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και δεν νομίζω ότι θα θέλαμε να διαγράψουμε μια θέση που ήδη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εγκρίνει. Εδώ δεν έχουμε λοιπόν μια ανάληψη υποχρέωσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και μόνο. Πρόκειται για μια πρόσκληση προς τις βιομηχανικές χώρες στις οποίες περιλαμβάνεται και η Κίνα και οι Ηνωμένε Πολιτείε και άλλες χώρες και οι χώρες κατοφλίου να κινηθούν προς την κατεύθυνση της επίτευξης αυτού του στόχου που ζητάει το πάνω για την κλιματική αλλαγή. Ο Πέτερ Λίζε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, <clears throat> πιστεύω, αντίθετα από άλλους συναδέλφους, ότι θα πρέπει το έργο του IPCC, του πάνω για την κλιματική αλλαγή, να είναι η βάση της εργασίας μας δεν νομίζω ότι αυτό σημαίνει ότι παραγνωρίζουμε άλλες απόψεις του Πάπα ή του Νταλάη Λάμα ή άλλων επιστημόνων. Εμείς είχαμε συζητήσει το θέμα αυτό και με τον πρόεδρο της ε, Επιτροπής αυτής την, ε, το Φεβρουάριο το Μάρτιο. Όλοι αυτοί οι οποίοι διαμφισβητούν αυτά τα οποία λέει το IPCC να επανέλθουν σε αυτό και θα έχουμε τον Νοέμβριο και πάλι και μια συζήτηση με τον αντιπρόεδρο αυτού του πάνελ. Δεύτερον, οι, έχουν δίκιο οι συνάδελφοι, 20% σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι η απόφασή μας και 30% εάν υπάρξει συμφωνία στην Κοπενχάγη. Αλλά είναι σωστό αυτό το οποίο είπε και ο πρόεδρος μας, ότι εάν θέλουμε να πετύχουμε μια διεθνή συμφωνία, θα πρέπει να κινηθούμε και μέσα στην ψαλίδα του 25 με 40%. Δεν είναι απαραίτητο να βρισκόμαστε στο άνω όριο. Η Ιαπωνία μετά από πολλές δυσκολίες έχει φτάσει σε μια απόφαση του 25%. Και οι Αμερικανοί μπορεί να μην περιοριστούν στο 25%. Επομένως υπάρχει η δυνατότητα να φτάσουμε σε ένα στόχο του 30%. Λοιπόν, αυτή είναι μια απόφαση η οποία πρέπει να ληφθεί στην Ολομέλεια. Αλλά είναι σωστό να περιέχεται αυτό το ερώτημα στην προφορική μας ερώτηση. Στην έκθεση Florence, στο σημείο 3, αναφέρεται ο στόχος του, της μείωσης κατά 25 με 40%. Επομένως είναι σωστό να περιλαμβάνεται και στην προφορική μας ερώτηση. Αλλά δεν λέει η έκθεση Florence ή κάποιο άλλο κείμενο ότι πρέπει να είμαστε ακριβώς στο 40%. Θα πρέπει να αφήσουμε ανοιχτό το θέμα του άνω άκρου της ψαλίδας. Θα πρέπει λοιπόν εμείς να καθορίσουμε τη στάση μας στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Ενδεχομένως χρειάζεται να υπάρξει και μια χωριστή ψηφοφορία για το αν θα πρέπει αυτό να περιληφθεί στο ψήφισμα τελικά ή όχι. Ευχαριστώ, λέω πρόεδρος. Αναφέρεστε στην έκθεση Φλόρενς της 4 Φεβρουαρίου του 2009 αλλά υπάρχει και η έκθεση χάση και το ψήφισμα της 11ης Μαρτίου 2009 όπου υπάρχει εκπεφρασμένα συνολική μείωση ε, εκπομπών θερμοκηπίου στο άνω όριο της ψαλίδας 25 με 40% όπως ε, προβλέπεται στην έκθεση αξιολόγησης του πάνελ για την κλιματική αλλαγή. Επομένως και αυτό είναι επίσημη θέση του Κοινοβουλίου. Το Μάρτιο υποστηρίξαμε το άνω άκρο της ψαλίδας. Εντάξει. Νομίζω ότι θα μπορούσε αυτό να κριθεί από μια ψηφοφορία. Το αν θα πρέπει να έχουμε αναφορά στο άνω άκρο ή, το, ή όχι της ψαλίδας. Εγώ νομίζω ότι εδώ είμαστε κάπως περιορισμένοι σε ό,τι αφορά την παρουσία και θα μπορούσαμε να δώσουμε μια λανθασμένη ε, εικόνα αντιπροσωπευτικότητας. Νομίζω ότι θα ήταν καλύτερο την επόμενη εβδομάδα να καταλήξουμε σε μια απόφαση και εσείς θα ήταν χρήσιμο να είμαστε πιο συνεπείς και να μην αλλάζουμε θέση κάθε μήνα. Και πάλι σας λέω ότι αυτή τη στιγμή θέτουμε αυτό τον αριθμό μέσα στα πλαίσια μιας ερώτησης και όχι στα πλαίσια μιας διατύπωσης απαιτήσεων. Θα ήθελα να σας προτείνω λοιπόν να δεχτούμε την διατύπωση αυτή όπως είναι αν υπάρχουν διαφορέ μπορούμε να το εξετάσουμε και πάλι την επόμενη εβδομάδα που θα υπάρχει πληρότερη σύνθεση τη επιτροπή μας. Λίζε, συμφωνεί ότι πρέπει να είμαστε συνεπείς και όχι ασυνεπείς και ασυνάρτητοι με τον εαυτό μας. Κύριε Ζέμπα, εγώ θα ήθελα να προτείνω πράγματι να αναβάλουμε την ε, απόφαση πρέπει να γίνει κάποια ψηφοφορία γιατί υπάρχουν διαφορετικές απόψεις για το θέμα αυτό και η αποφασιστική λοιπόν απόφαση πρέπει να ληφθεί επί τη βάση της ε, έκθεσης Florence. Νομίζω ότι θα πρέπει λοιπόν να επανέλθουμε σε αυτό το θέμα και να αποφασίσουμε για τη συμπερίληψη του ποσοστού αυτού σε μια χωριστή ψηφοφορία. Αυτό θα ήταν το πιο πρόσφορο για να φανεί η άποψη της Επιτροπής μας. Κυρία Χάση. Uh, Κοιτάξτε. Ναι, να αναβάλουμε την ψηφοφορία, αλλά εάν ψηφίσουμε σήμερα, να μην ξεχνάμε ότι ακόμα και ένα μέλος μπορεί να διαφωνήσει μια προφορική τροπολογία στην προφορική ερώτηση. Äh, μία τροπολογία μπορεί να αντιμετωπίσει αυτή την αντίρρηση ο προϊόν μέλους. Είναι γεγονός, αλλά όχι μία χωριστή ψηφοφορία όταν ζητηθει λέει ο προεδρο Έτσι μου είπε <laughs> έτσι λέει ο πρώην πρόεδρο της Επιτροπής ε, Κανονισμού. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν μία αίτηση για χωριστή ψηφοφορία για το άνω άκρο τη ψαλίδας. Ωραία. Ψηφίσουμε τότε ποιος υποστηρίζει να συμπεριληφθεί στην ερώτηση να μην συμπεριληφθεί μάλλον το άνω άκρο στην προφορική ερώτηση. Ποιος είναι υπέρ αυτού, να μην περιληφθεί. Ναι ναι, Είναι okay. The 12. Ποιος είναι εναντίον της διαγραφής. Αποχές. Ο, ούτε ο Καλ Φλόρενς θα μπορούσε να το αλλάξει αυτό. Παραμένει λοιπόν και επομένως ποιος είναι υπέρ του να τεθεί το ερώτημα αυτό στην Κομισιόν με αυτή τη μορφή. Ψήφι υπέρ. Κατά. Ωραία. Αποχές